σιγά να ξεκινάμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να κηρύξουμε την έναρξη τώρα της ακρόασης για το θόρυβο. Σας καλωσορίζω όλους θερμότατα ιδιαίτερα όλη αυτή είναι τίτλο. Ε, την Υφυπουργό του Πολωνικού Υπουργείου Μεταφορών. Καλώς ορίσατε. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πρόβλημα ιδιαίτερο η χορύπανση και ο θόρυβος και πρέπει να λυθεί για να έχει μέλλον και η κινητικότητα. Και αυτό αφορά και τον αυτοκινητόδρομο και το σιδηρόδρομο. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ε, έχουμε πολύ καλούς προσκεκλημένους σήμερα επισκέπτες. Ε, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την παρουσία τους το πρώτο πάνελ ε, απαρτίζουν ο κύριος Μπένχαρτ Μπέργκερ στη Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος και ο Μάρκ Βίτλ από το Κέντρο Στρατηγικής και ε, Υπηρεσία Αξιολόγησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλώς ορίσατε. Για δέκα λεπτά θα λάβετε το λόγο. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει από σας, παρακαλώ. Honorable members of Parliament, ladies and gentlemen, Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας, για το θόρυβο και τη σχετική οδηγία, αλλά και για τη διοργάνωση της παρούσης ακρόασης. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε κιόλας. Ε, είναι μεγάλη χαρά για μένα, ευκαιρία που έχω να σας μιλώ, για το που βρισκόμαστε με την αξιολόγηση της οδηγίας για το θόρυβο και γενικότερα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντο πρόσφατα εξέδωσε μια έκθεση που λέγεται «Θόρυβο στην Ευρώπη το 2014» και δείχνει ότι η οδική κυκλοφορία είναι η πιο ρηπογόνο από πλευρά ηχορύπανση. 125 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου ε, υφίστανται τι ε, συνέπειες του θορύβου, ενοχλούνται από το θόρυβο αυτό. Ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, διότι η εφαρμογή της οδηγίας έχει καθυστερήσει. Οπότε τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα έτσι χαμηλότερα από την πραγματικότητα. 30 με 50 χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις ε, πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο θόρυβος επηρεάζει πάρα πολύ ανητικά άσχημα την υγεία των ανθρώπων και ο δεύτερος μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος μετά την ύπαρση την ατμοσφαιρική. Η χορύπανση όμως δεν επηρεάζει μόνο την ε, ανθρώπινη υγεία έμεσα, αλλά και άμεσα. Είναι βάρος για το σύστημα υγείας, προκαλείται ε, απώλεια παραγωγικότητας, άρα και πρόβλημα στις ευρωπαϊκές οικονομίες. In of ε, συνέπεια όλων αυτών λοιπόν ποια είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον μέχρι το 2020 έχει δεσμευτεί να μειώσει σημαντικά την ηχορύπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσει πιο κοντά στα επίπεδα που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και αυτό είναι αυτολεξία αυτό που αναγράφεται ε, στο πρόγραμμα. Και τώρα σε λεπτομέρειες χρειαζόμαστε μια πολιτική για την ηχορύπανση που να είναι ε, ενημερωμένη με βάση τα τελευταία δεδομένα και χρειαζόμαστε μέτρα για να μειώσουμε το θόρυβο στην πηγή και επίσης να ε, βελτιώσουμε την πολεοδομία και την, το σχεδιασμό των πόλεων. Το πρόβλημα του θορύβου είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών μελών χρειάζεται ε, να ενέχονται και οι περιφερειακές αρχές και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ που μιλώ εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο βασικούς στόχου. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε στο, το θόρυβο στην πηγή, ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με βάση το πώς σχεδιάζουμε τους δρόμους μας. Υπάρχει μια οδηγία λοιπόν για τον περιβαλλοντικό θόρυβο που καλύπτεται στο γράμμα. Ε, τι στόχο έχει όμως τώρα. Να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση έτσι ώστε να αποφύγουμε ή να προλαμβάνουμε ή να μειώνουμε ε, την έκθεση, τον κίνδυνο για την υγεία που προκαλείται από έκθεση σε θόρυβο. Για να γίνει αυτό η οδηγία έχει διτή προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα συλλέγονται στοιχεία για την έκθεση στο θόρυβο και χρησιμοποιούνται αυτά έτσι ώστε ε, οι πάντες να είναι ενήμεροι για το πώς έχει ε, ο θόρυβος ε, στην πηγή, καταγράφεται δηλαδή η πηγή του θορύβου. Άλλο σημαντικό στοιχείο της οδηγίας είναι ότι επιμένει στην δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια δράσης, έτσι ώστε να μετριαστεί το πρόβλημα. Αυτό το γράφει η ίδια οδηγία, είναι κατοχυρωμένη η δημόσια διαβούλευση στην οδηγία. Τι δεν κάνει η οδηγία, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό ξεκάθαρα. Δεν βάζει οριακές τιμέ. ούτε στόχους, ούτε τίποτα τέτοιο ποσοτικό, ούτε ορίζει ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά είναι θέματα δικά του. Για να συλλέξουμε λοιπόν στοιχεία ε, ακριβή, συνεπή και συγκρίσιμα για την έκθεση σε θόρυβο, θα πρέπει οι μέθοδοι να είναι παρόμοιε, αντίστοιχε. Προφανώ, γιατί αν μετράς με διαφορετικέ μεθόδου, δεν είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματά σου. Γι' αυτό μεγάλο βήμα προ τα εμπρό έγινε το 2015. Συμφωνήθηκε μια νέα κοινή μέθοδο ε, για την εκτίμηση του θορύβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το παράρτημα 2. Και η μέθοδο λέγεται κνοσό. Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πώς το μετράμε. Ε, με διάφορους τρόπους ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Στόχος ε, του παραρτήματος 3 είναι και πάλι να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Έχει αρχίσει μια προκαταρκτική εργασία ήδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά τις εργασίες του ΠΟΗ, του τομέα Ευρώπη για να ε, προχωρήσουμε και να συγκρίνουμε τα δικά μας στοιχεία και να τα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη ως κατευθυντήρες γραμμές. Παράλληλα με την εκπόνηση αυτής της οδηγίας στο παράρτημα 2 και 3, αυτό τον καιρό αξιολογείται ε, και στο πρόγραμμα REFIT τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το ξέρετε, που αξιολογεί την κείμενη νομοθεσία ως προς την αποτελεσματικότητα. Έχουμε δει τι πρωτοβουλίε έχουν ληφθεί και έχουν εφαρμοστεί εδώ και καιρό για να ε, μετρηθεί και να αξιολογηθεί η επίδοση συγκρινόμενη με κάποια στάνταρ κριτήρια, προδιαγραφές. Αυτά τα κριτήρια τα βλέπετε στην παρούσα διαφάνεια. Θα πρέπει η αξιολόγηση να κοιτάξει αν οι στόχοι της οδηγίας ε, έχουν ε, αποδόση είναι ικανοποιητική, δηλαδή αυτό έχει να κάνει το, κόστος, την ωφέλεια και το διοικητικό άκθος. Επίσης, κοιτάει η αξιολόγηση αν είναι συνεπής με άλλη νομοθεσία η οδηγία αυτή, αν είναι ενισχύει ε, η στόχη και αν ε, υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν από μόνα τους τα κράτη-μέλη. Έχουμε ένα στοιχείο λοιπόν ευρωπαϊκής υπεραξίας. Guidelines of the European Commission on the Refit Program, we have published the roadmap. ένα οδικό χάρτη ε, έχουμε δημοσιεύσει το Νοέμβριο του 2015. Μπορείτε να το βρείτε ε, στη ε, ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταλάβετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα διάφορα στοιχεία. Έχουμε ζητήσει, έχουμε αναθέσει μια μελέτη σε ένα εξωτερικό συνεργάτη, γιατί αυτό πρέπει εξωτερικός να το κάνει, που κάθεται εδώ εκ δεξιών μου, και βασίστηκε ε, σε πάρα πολλά στοιχεία, ε, ενημέρωση, πληροφορίες, απόψεις των ενεχομένων και θα εξηγήσει ε, μετά τη μελέτη που θα αποτελέσει τη βάση για τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση ε, θα λάβει μορφή εγγράφου εργασίας, εσωτερικό, έτσι ήθιστε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα καταλάβετε ότι δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή για τα ευρήματα, για την ουσία. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τα ευρήματα της μελέτης, που είναι σημαντική βάση, θα πρέπει να δούμε και κάποια επιμέρους στοιχεία, που είναι η δημόσια διαβούλευση, που έγινε αρχές του έτους και επίσης θα πρέπει να ε, συμβουλευτούμε και τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επίτροπης. Άρα μπορεί να καταλήξουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα ε, με τον ε, συντάκτη της μελέτης, αλλά θα τα δημοσιεύσουμε και τα δύο για λόγους διαφάνειας ταυτόχρονα. Η επόμενη έκθεση εφαρμογής που προβλέπεται από την ίδια την οδηγία θα κατατεθεί το 2017 και πάλι θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ε, στην έκβαση της μελέτης για την ε, υλοποίηση και την ε, εκτέλεση της οδηγίας αυτής και θα δίνει και μια επισκόπηση του ακουστικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με το αποτέλεσμα θα έρθει αυτή η έκθεση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στι αρχές του 2017 και ενδεχομένω να προβλέπει και νέα μέτρα ή νέα βήματα για την πολιτική κατά του θορύβου. Συνοψίζω. Έχουμε μια μέθοδο εκτίμησης του θορύβου και θα πρέπει τα κράτη-μέλη από το 2018 και μετά να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο συνεργαζόμαστε με τον τομέα Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα κράτη-μέλη. Προγραμματίζουμε την έκθεση αξιολόγησης με βάση την εξωτερική μελέτη να την καταθέσουμε μέχρι τα τέλη του έτους. Και τέλος, μια δεύτερη έκθεση ε, εφαρμογής προβλέπεται για την αρχή του 2017 και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και νέα μέτρα για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την καταπληκτική τήρηση του χρόνου. Αυτή ήταν η πρώτη ομιλία. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μακ Γουίτλ ε, να μας παρουσιάσει τη μελέτη. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Μπέργκερ, πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι ευρωβουλευτές, και κύριοι. Είμαι ο Μάικ Χουίτλ από το Κέντρο Στατηγικών Ερευνών και Αξιολογήσεων και κάναμε την αξιολόγηση της οδηγίας για, το, για την ηχορύπανση χρησιμοποιώντας τη βοήθεια περιβαλλοντικών οικονομολόγων και οτορινοραλικολόγων ειδικών στα θέματα αυτά. για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αναχέτησης της συγχωρήπανσης όπως προέκυπταν από την οδηγία αυτή. Θέλω να σας παρουσιάσω κατευθείαν τα πορίσματα αυτής της μελέτης. Δύο ήταν οι βασικές μας μέρημνες, όπως είπε ο κ. Μπέργκερ. Πρώτα απ' όλα οι απαιτήσει της οδηγίας να εκπονείται πενταετής ε, επισκόπηση της ολυλοποίησης των βασικών νομοθετικών διτάξεων της οδηγίας για να δούμε αν ήταν αν υπήρχαν θέματα υλοποίησης, προβλήματα μέσα σε μια συγκεκριμένη πενταετία. Και κατά δεύτερον, να αποτιμηθεί η οδηγία στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT επισκόπησης μαζί με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής και τις σχετικές αναθεωρήσεις της θα δημοσιευτούν στο τέλος της χρονιάς. Ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, απλώς να πω ότι ήταν μια αυστηρότατη μεθοδολογία. Στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων είχαμε πάνω από 100 συμμετοχές με σχετικά εργαστήρια, με γραπτές συνεισφορές και διαρκή ε, διάλογο με τους ενδιαφερομένους κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης. Να προχωρήσω στα θέματα της αξιολόγησης. Αυτά καλύφθηκαν στην προηγούμενη παρουσίαση, αλλά επί της ουσίας πρέπει να δούμε τα κλασικά θέματα αξιολόγησης, που μια ανεξάρτητη αξιολόγηση καλύπτει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα οποία έπρεπε εδώ να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες της οδηγίας για την χορύπανση. Να σας δείξω μερικά από τα πορίσματα για καθένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης. Για το κατά πόσο ήταν εύστοχη η οδηγία λοιπόν. Μια κοινή προσέγγιση στην αποτίμηση του περιβαλλοντικού θορύβου της συγχωρήπανσης είναι ένας ε, εύστοχος, ε, μια προτεραιότητα σκόπιμη, γιατί επιτρέπει στα κρατημέλη να κινηθούν προς μια κοινή προσέγγιση για την ε, συγκέντρωση δεδομένων. Αυτό επί σειρά ετών και με πολύ τεχνική δουλειά, για να υπάρξει μια κοινή μεθοδολογία αποτίμησης μέσω του συστήματος γνωσός. Ο στόχος αυτός καθεαυτός είναι ένας στόχος ενδιάμεσος βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κατά πόσον ε, ωφελεί σε κάτι. Να υπάρξει ίσως ένας στόχος που να ευνοεί τη δημόσια υγεία ώστε να ε, επαληθεύουμε το τι επιτυγχάνει μακροπρόθεσμα η οδηγία. Η κοινή προσέγγιση θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να διαμορφωθεί. Και είναι σίγουρα ένα ενδιάμεσο βήμα προς τον απότερο στόχο, τη βελτίωση τη διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και την ε, μείωση τη συγχωρήπανση ή των επιπτώσεων της στην υγεία. Ω προ τον δεύτερο στόχο, την νομοθεσία που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή αυτή τη οδηγία ήταν πραγματικά εύστοχη, διότι ο ρόλο της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, την χορύπανση, ήταν να ασχοληθεί με το θόρυβο στην φάση του δέκτη. Ενώ η οδηγία για τις πηγές του θορύβου ασχολείται με το θόρυβο αναπηγή παραγωγής του, ένα είδος μεταφοράς και ανασυγκεκριμένα περιβάλλοντα. Εκεί χρειάζεται να συσχετίσουμε τις πηγές του θορύβου με το τοπικό επίπεδο θορύβου και τη συχνότητα. Ας περάσουμε τώρα στην συνοχή, την συνεκτικότητα μάλλον της οδηγίας. Σε επίπεδο νομικού κειμένου υπάρχουν λεπτομέρειες στους ορισμούς ε, και κοιτάξαμε κατά πόσον τα άρθρα μεταξύ τους ε, συνδυάζονται σωστά. Η οδηγία ε, στο κείμενό της λοιπόν είναι γενικώ συνεκτική, όμως σε κάποια σημεία η διατύπωση του νομικού κειμένου θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί. Όπως κάποιες φορές οι ορισμοί σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήξαμε ότι οι ευθύνες των κρατών μελών είναι μάλλον σαφείς για τους περισσότερους ενδιαφερομένους, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχει και σύγχυση για το κατά πόσο μερικά μέτρα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στα προγράμματα αντιμετώπιση τη συγχωρήπανση ή όχι. Επίσης, το κατά πόσον ο ορισμός σιωπηλών αθόρυβων περιοχών είναι υποχρεωτικός ή όχι. Αυτά δεν ήταν τελείως σαφή από την οδηγία και το κείμενό της και μόνο. Ως προς την ε, εξωτερική συνοχή, δηλαδή το κατά πόσον η οδηγία για την χορύπανση και άλλη σχετική νομοθεσία, κυρίως η οδηγία για τις πηγές του ρήβου, μπορούν να συνδυαστούν, εκεί καταλήξαμε ότι οι διαφορετικές μορφές νομοθεσίας αλληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή αυτή η οδηγία είναι το μόνο νομοθέτημα που απαιτεί να υπάρξει χαρτογράφηση του σχεδιασμού του, του, ίδιου του θορύβου ε, καθώς και συγκεκριμένα προγράμματα δράσης σε τοπικό επίπεδο. Ως προς το εύρος, τον, την υγεία δηλαδή της, ε, του νομοθετήματος έπρεπε να δούμε κατά πόσον σε σύγκριση με άλλα νομοθετήματα μπορεί να σταθεί αυτή η οδηγία Δύο μόνο ενδιαφερόμενοι εντόπισαν προβλήματα σε σχέση με τον ε, βιομηχανικό θόρυβο, μεγάλης κλίμακας δηλαδή, σε σχέση με την οδηγία ε, END και την οδηγία για, την, ε, για τον βιομηχανικό θόρυβο. Εκεί τα πράγματα και τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Και τα κράτη-μέλη, μόνο σε μερικά κράτη-μέλη εντοπίστηκαν προβλήματα βάσει των πληροφοριών των ενδιαφερομένων ως προς την αποτελεσματικότητα. Συνολικά είδαμε ότι έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδος προς το να διαμορφωθεί μια κοινή προσέγγιση. Η σημασία αυτής πρέπει να τονιστεί, ιδίως εφόσον η οδηγία εγκρίθηκε τη στιγμή που μόλις τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν κάποια νομοθεσία περί χορύπανσης και ήταν μάλιστα και πολύ αποκλίνουσες οι προσεγγίσεις τους ως προς τις μεθόδους συμπίλησης ή τον τρόπο που μετρά, μετρούσαν την έκθεση στον θόρυβο. Θα χρειαστεί καιρό για να συνδυαστούν όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όπως είπε ο κύριος Μπέργκερ, ιδιαίτερος η δημιουργία του συστήματος Κνωσός από το 2007 στο 2015 και που οδήγησε στην έγκριση της κοινή οδηγίας της Επιτροπής για την ε, μεθοδολογία των αξιολογήσεων είναι ένα μείζον βήμα για την κοινή προσέγγιση. Για να ορίσουμε τις σχέσεις αξιολόγησης και τους λόγους μεταξύ της έκθεσης και των επιπτώσεων στην υγεία υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά περιμένουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναθεωρήθηκαν, καθώς και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που επηρεάζονται από αυτή τη δημοσίευση. Ω προ το δεύτερο στόχο, δηλαδή την επικαιροποίηση τη ε, νομοθεσία που βρίσκεται στην πηγή, εκεί η εικόνα είναι κάπω πιο συγκεχημένη, πιο μεικτή. Από τη μια έχει επιτελεστεί πρόοδος ως προς την ως προς τον σχεδιασμό πολιτικής μέσα από τομείς προτεραιότητας και καθώς η οδηγία αυτή είναι ένα σημαντικό στρατηγικό σημείο αναφέρεται ένα από τα εργαλεία, η μελέτη αντικτύπου, στο, σε μια από τις σκέψεις. Αυτό έχει να κάνει και με την νομοθεσία φυγή. Όμως, τα δεδομένα για την έκθεση του πληθυσμού δεν έχουν χρησιμοποιεί ακόμη όσο διεξοδικά θα έπρεπε. Τόσο διεξοδικά μάλλον όσο θα έπρεπε. Και αυτό έχει να κάνει και με τις καθυστερήσεις των κατώμελών μελών στην υποβολή των στοιχείων. Και υπάρχουν και προβλήματα συγκρισιμότητας. Στι διάφορε φάσει τη υλοποίηση και σε σχέση με τα δεδομένα έκθεση στην χωρίπαψη. Στο μέλλον πάντω, τα δεδομένα αυτά και εφόσον ε, συμπληρωθούν και είναι πιο πλήρη και πιο συγκρίσιμα θα επιτρέπουν να ενισχυθούν οι αμόψεις μας, όπως από, κάποιες, ε, από αυτά που προκύπτουν από κάποιες σχετικές δημοσιεύσεις. ως προς τις λεπτομερέστερες, ε, στα λεπτομερέστερα συμπεράσματά μας για την αποτελεσματικότητα, υπάρχει θέμα με, την, ε, με το κατά πόσο είναι πλήρη τα δεδομένα. Είδαμε στις φάσεις 1 και 2 να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις από την υποβολή των στοιχείων των μελών. Και αυτό απηχεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί από κάτω μέλος σε κάτω μέλος. Κάποιες χώρες έχουν τελείως αποκεντρωμένη προσέγγιση με τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών φορέων και ενδιαφερομένων. Υπάρχει πρόβλημα έλλειψη πόρων πολλέ φορέ, κυρίω λόγω τη χρηματοοικονομική κρίση. Και συνολικά βλέπουμε ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα, αλλά υπάρχει και ανάγκη κοινή προσαγγίση να ενισχυθεί ω προ την εθνική εφαρμογή των μέτρων. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις έχουμε τώρα ή σύντομα σχόλια, εν πάση περιπτώσει. Ο Βίμ Φαντενκάμ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε ακουστικά, παρακαλώ. Connecting Europe είναι αυτό. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις έχω προς τον κύριο Μπέργκερ. Τον άκουσα να λέει ότι ο αυτοκινητόδρομος παράγει περισσότερο θόρυβο από ότι τα τρένα. Αυτό δεν είπατε ότι ε, και σε σύγκριση με τα τρένα είναι πιο θορυβόδης η κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους. Δεύτερη ερώτηση. Άκουσα να λέτε ότι 30 με 50 χιλιάδες είναι λέει πρόοροι θάνατοι ετησίως έτσι που βασίζονται στο θόρυβο. Ε, λόγω του θορύβου. Αυτό τώρα πώς το μετράτε. Πώς πεθαίνει από θόρυβο, κουφέρεσαι. δηλαδή, πώς πεθαίνει από το θόρυβο. Ε, ε, αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο να επεκταθείτε. Και ε, η οδηγία αυτή είναι του 2002. Τώρα θα φέρετε καμιά αναθεώρηση ή προσπαθείτε να εφαρμόζετε σωστά αυτή η οδηγία. Αυτές ήταν οι τρεις ερωτήσεις προς τον κύριο Μπέργκερ. Ευχαριστώ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Πολλές είναι οι ερωτήσεις που θα είχα να κάνω για το θόρυβο και πολύ μεγάλη φασαρία γίνεται στα κράτη-μέλη ε, και εκνευρισμός υπάρχει και για την αναέρια κυκλοφορία και για το σιδηρόδρομο το θέμα δεν είναι ότι δεν έχει δραστηριοποιηθεί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω και πάλι στα πλαίσια της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη ε, έχουμε ελευθερώσει κονδύλια για την ανανέωση του τροχαίου υλικού ε, στο σιδηρόδρομο. Αλλά αυτά ήταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα έχουμε μια τρέχουσα περίοδο η οποία σχεδόν έχει περάσει το μισό της θητείας μας. Ε, ωραίες οι διαπιστώσεις, αλλά προς το πού θέλουμε να πάμε. Μου λείπει λίγο η κατεύθυνση. Ωραία αυτά που μας λέτε, αλλά πού το πάμε. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα χάσμα. Ανατολής Δύσης, αν το πω έτσι. Βεβαίως η Γερμανία έχει τα περισσότερα βαγόνια να κυκλοφορούν στο σιδηρόδρομο, αλλά μπορεί εύλογα να πει κάποιος ότι η Γερμανία τα πάει καλά από ανανέωση του τροχαίου υλικού ως προς τα αθόρυβα βαγόνια. Αλλά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν με την ίδια ταχύτητα. Οπότε, πώς να το πω τώρα, ε, κάνουμε μισές δουλειές, δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό. Και ε, έχω ρωτήσει και την Επίτροπο, την ίδια την κυρία Μπολτς μήπως θα είχε νόημα εκείνα τα κράτη-μέλη ε, που δεν προχωρούν να έχουν ένα κίνητρο, να έχουν ένα πριμ απόσυρσης, αν αποσύρουν τα παλιά βαγόνια και τα αντικαταστήσουν με νέο τροχαίο υλικό. Πώς το βλέπετε αυτό και τι προβλέπετε, τι φανταζεστε ε, τώρα τι προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν προγραμματίζει νομοθετικά μέτρα. Γιατί σχεδόν δυόμιση χρόνια έχουν περάσει από τούτη εδώ τη θητεία και το θέμα του θορύβου είναι Πολύ υπαθώ. Είναι ένας εκνευρισμός μόνιμος και μια φασαρία και το πολιτικό επίπεδο τι κάνει για τους ανθρώπους. Τουλάχιστον οι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητά τους ότι κάτι κάνεις για να το αντιμετωπίσει. Και αν ασφάλω παρακαλώ μην διστάσετε να με διορθώσετε. Ευχαριστώ Τζάκη Φώστερ. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να διορθώσουμε αυτή την ακρόαση σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ξέρω πως ο πρόεδρος ε, κατοικεί σε μια περιοχή όπου υπάρχει φοβερή χορύπανση από τα τρένα. Γνωρίζω πολύ καλά πως ο θόρυβος είναι κάτι δεν ενοχλητικό. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπος μετριασμού. Νομίζω ότι τα πάμε καλά στην Ευρώπη σχετικά και πολλά κράτη προσπαθούν να βρουν τεχνολογικές λύσεις για την επίλυση του προβλήματος. Πολύ καλά κάνουμε και έχουμε οδηγία για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση των 21ου αιώνα. Έχουμε κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε κάποια ζητήματα ειδικά εμεί εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Θυμάμαι ότι ήμουν μέλος τη Επιτροπής Μεταφορών πριν από αρκετό καιρό όταν μιλούσαμε για το θέμα των, ε, του πετρελαίου που χρησιμοποιούν τα σκάφη, τα πλοία διότι θυμόμουν ότι πολλές γυναίκες έχασαν ε, τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους επειδή κατοικούσαν κοντά σε ε, λιμάνια ή σε ποτάμια τα οποία, τα οποία κινούν τα πλοία που χρησιμοποιούσαν ε, κάψιμα υψηλή περιοχτικά δαθείου. Θυμάμαι και τον συνάδελφο Ινβανεκάμπ μια παρουσίαση που είχε κάνει. Και εσείς κύριε Μπέργκερ είπατε ότι μεταξύ 20 και μάλλον μέχρι 30 και 50 χιλιάδων ανθρώπων χάνουν τη ζωή του ετησίω λόγω του θορύβου. Ποια είναι αυτά τα άτομα, πού κατοικούν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, δεν ξέρω, έχουν εκδοθεί ε, πιστοποιητικά θανάτου ότι ε, ο θάνατος οφείλεται στην ε, τη χορύπανση. Υπάρχουν στοιχεία για το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία δεν έχουν καν κάποιες διαδικασίες για να μπάνουν παρόμοια στοιχεία. Λοιπόν, βασίζεται ενδεχόμενα σε, σε λίγα κράτη. Μπορείτε να μας φέρετε όμως κάποια στοιχεία και όχι μόνο υποθέσεις ότι κάποιος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του από την χορύπανση. Πρέπει να τα στάσουμε σε βάθος τα θέματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως ενήλικες που θέλουν να προοδεύσουν, να προχωρήσουν, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο πραγματικό. Δεν ζούμε σε έναν πλασματικό κόσμο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στοιχεία για να μου καλύψετε και τις ανησυχίες μου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ανάμεσά μα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Ντομινίκ ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω στο θέμα που έθεσε ο Βίν και ο Ζάκη ως ε, γιατρός ε, θα με ενδιαφέρει η ποιότητα του ήχου. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι ο ήχος προκαλεί ε, άγχος, στρες και ως εκ τούτου μπορεί να προκαλέσει ε, φυσιοπαθολογικές καταστάσεις, αρνητικές. Τώρα για θανατηφόρους το αμφιβάλλω. Έχω κάποια ερωτηματικά αν και ότι γνωρίζω ότι μπορεί να συμμετάσχει στην πρόκληση κάποιες παθολογίες. Εντάξει, ο θόρυβος δεν ε, οδηγεί στο θάνατο, εκτός περιπτώσει, περιπτώσεις, αλλά εντάξει, αν είσαι James Bond, αλλά με εκπλήσουν λοιπόν αυτό το, αυτές οι 30 50000 ε, άτομα τα οποία χάνουν τη ζωή τους ε, από την χορύπανση. Θεωρώ λοιπόν να μιλήσουμε για θανάτους με αιτία των θόρυβων, δεν μπορεί να είμαστε αξιόπιστοι. Τώρα, αν συμμετέχει στο 15% σε 150.000 θανάτου, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Πρόκειται για μια μελέτη εξάλλου, η οποία είναι μια μελέτη ποσοτικής φυσή, Θα ήθελα να ε, ε, βάλουμε την έννοια τη ποιοτική έκθεσης. Ο, ο θόρυβος είναι μια συγνότητα. και ο επιθετικός χαρακτήρας, ε, το επίπεδο ανοχής και τα ε, παράγοντα και παράγοντες είναι ε, επίση κάτι το σημαντικό. Κοιτάξτε, υπάρχουν τόροι που, είναι, που, δεν ακούγονται καν. Είναι, δεν είναι πάντα θέμα δεσιμπέλο θόρυβος και ανάλογα με την πηγή η οποία εκπέμπει τον θόρυβο. Μπορούμε να έχουμε λευκό θόρυβο, ο οποίο ε, μπορεί να έχει πολύ ψηλό ποσοστό δεσιμέλ. Ε, εξαρτάται λοιπόν από τον ποσοστό της, ε, από την συχνότητα, συγγνώμη. Παρακαλώ μιλήστε, μιλήστε μας για την ε, ποιότητα του ήχου και αναφερθείτε στην πηγή, διότι ο ήχος ε, του σιδηρόδρομου δεν είναι ο ίδιος με το, αυτός τον δρόμου και αυτός που ε, προκαλείται σε ένα αεροδρόμιο. Ένα αεροπλάνο το οποίο απογειώνεται δεν δημιουργεί την ίδια δεσιμπέλ με έναν αυτοκινητόδρομο. Και τέλος, πέραν από ε, τα θέματα του εντοπισμού θα πρέπει να ε, εξετάσουμε το πώς μπορούμε να διορθώσουμε ε, το, το θόρυβο. Τώρα, αν είναι να τον εξαφανίσουμε, να τον απαλύσουμε τον θόρυβο, αυτό είναι μάλλον αδύνατον. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές ε, που, μέσω των οποίων δημιουργούμε αντίμετρα οι λύσει ε, δεν είναι πάντα τόσο προφανεί από πολιτική σκοπιά και η τεχνική έννοια του θορύβου και η ε, τεχνολογική της, ε, της του θορύβου νομίζω ότι αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με τρόπους διαφορετικούς σε πολιτικό επίπεδο. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Λιουκασεύσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Μιλήσατε για πολλές χιλιάδες ε, θανάτους. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω σε τι βασίζεστε, γιατί από ό,τι, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία αναφορικά με τις επιπτώσεις της συγχωρήπανσης επί της υγείας. Και μία ερώτηση τώρα για τον κύριο Μπέργκερ. Το να μειωθεί ε, ο θόρυβος, η χορύπανση, αυτό ε, επιφέρει ένα τεράστιο κόστος. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν έχετε εκτιμήσει, έχετε αξιολογήσει το, το κόστος και ε, με ποιο τρόπο μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτέ οι προσπάθειε. Είπατε επίση ότι η οδηγία που επεξεργάζεστε δεν θα προβλέπει κάποια ρύθμιση ή κάποια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου θα θέλω να μάθω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επιβάλλει υποχρέωση για τον εξυγχρονισμό των ε, τρένων των εμπορικών και ή όλα θα εξαρτηθούν από την απόφαση των επιμέρους κρατών μελών. Διότι όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, το κόστος είναι τεράστιο και η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από κράτος σε κράτος. Η κατάσταση έχει διαφορετικά σε μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης από ότι σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Στην Πολωνία, παραδείγματος χάρη, τα βαγόνια έχουν ρόδες ε, ε, μονομπλοκ. Το κόστος λοιπόν θα είναι πολύ ψηλότερο από το κόστος το οποίο θα απαιτήσει μια αλλαγή στα, στους σειρμούς ε, της Δυτικής Ευρώπης. Ε, και τέλος θα ήθελα να μάθω εάν στην οδηγία θα την υπόψη και το επίπεδο της πυκνοκατοικίας, πυκνοκατοίκησης. Διότι ο, μεταφορές οι οδικές ή οι σιδηροδρομικές είναι πολύ διαφορετικές όπου η οι ειναι πολυ διαφορετικέ οπου η πυκνοτητα π.χ. στην Ολλανδία είναι τέσσερις φορές ψηλότερη από ό,τι στην Πολωνία. Και επίσης παίζει ρόλο κατά πόσο οι τροχές, ε, οι σιδηροτροχές παίρνουν ε, μέσα από πόλη ή όχι, όπως και οι αυτοκινητόδρομοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, Γεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν με είδατε προηγουμένω. ε. Συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Εντάξει. Έλεγα ότι οι συντονιστέ παίρνουν αυτόματα το λόγο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Πολλά υπόθηκαν ήδη για τα, τους θανάτους. Ε, μας φαίνεται λίγο μυστήριο, λίγο περίεργο και ο συνάδελφος Ντομινίκ Ρικέ είναι γιατρός, το απάντησε ε, αυτό με το άγχος που δημιουργείται μπορεί να προκληθούν θάνατοι. Βεβαίως, ε, θόρυβος έχει μεγάλη σχέση με τις μεταφορές και κάτι πρέπει να κάνουμε. Το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος ανυπόμονος γενικά, από το 2002 ότι λιβανίζουμε αυτή την οδηγία, τι θα γίνει. Και μαζεύεται στοιχεία. Ωραία, από το 2002 έχετε κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμιά διάσκεψη για το θόρυβο, όπως κάνουμε τώρα εμείς εδώ την ακρόαση αυτή. Από το 2002, ε, δεν τα έχετε μετρήσει πια, δεν, δεν, δεν, ξέρετε, κάτι δεν έπρεπε να έχει γίνει από τότε. Το ξέρω ότι είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών, γιατί υπάρχουν ε, αυτά ε, τα πανώ στους αυτοκινητοδρόμους, ε, προστατευτικές ε, τέτοιες υποδομές. Υπάρχουν και άλλα θέματα με τα καύσιμα, διακυροζίνη, να χρησιμοποιείται ηλεκτρισμός ή ακόμα και στα, στα αεροπλάνα ή κάποια συστήματα θόρυβης πέδησης. Το ξέρω ότι εσείς δεν κάνετε θαύματα, αλλά η χορύπανση είναι ρήπανση ε, του περιβάλλοντος και επηρεάζει το σύνολο περιβάλλον. Ε, εμένα αυτό με ανησυχεί κάπως και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούν να γίνουν περισσότερα και δεν μπορούν να γίνουν ταχύτερα από το 2002. Σας είπα τι με ανυπόμονη. Γιατί ε, το να κάνεις μόνο υποδομές σιδηροδρόμου στη Γερμανία σταματάει αυτό γιατί ο κόσμος λέει δεν θέλω τρένο, κάνει τόση φασαρία, δεν μπορώ τόσο θόρυβο. Άρα και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να καταπολεμηθεί η αιτία του θορύβου. Και σε όλες τις πολιτικές μεταφορών που ασκούμε θα πρέπει να έρθει πιο κοντά στο επίκεντρο της προσοχής και οικονομικά. Ο Μπέτερ Λούντκρεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους, την Τζάκι Φώστερ, τον Ντομινίκ Ρικέ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο πια να έχουμε τόσους νεκρούς από το θόρυβο. 50.000 είναι ένας αριθμός που συχνά χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως και οι συνάδελφοι πιστεύω και εγώ ότι χρειαζόμαστε λίγο καλύτερα στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία για να πιστούμε. Υπάρχει και το θέμα των συνθέτων υλικών ε, που συζητούσαμε και το πρωί, όπως έλεγε η συνάδελφος από την ε, Φιλανδία. Τα σύνθετα υλικά και τα συστήματα πέβησης ε, εξαιτίας της έλλειψης θερμότητας και την τον αντι... τις επιπτώσεις που έχουν οι χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ένα θέμα στη Ρωσία. Χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα, σύνθετα υλικά και εκεί, αλλά φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα τα φρένα των τρένων. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπω χρησιμοποιούμε λάθο τεχνικέ εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω δεν λειτουργούν απλώ. Μήπω να τα ξαναδούμε. Μήπω να κοιτάξουμε καλύτερα το ρωσικό παράδειγμα. Εάν είναι σε θέση τα δικά του τα συστήματα πέδηση να λειτουργούν καλύτερα, Ας προβλέψουμε κι εμείς ε, κανόνες που να μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όπως έλεγα λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία. Ε, θα πρέπει να πω ότι Καταλαβαίνω στην καθημερινότητα πως όλα αυτά μπορεί να δημιουργούν προβλήματα, αλλά θα ήθελα κάτι λίγο πιο χειροπιαστό, λίγο πιο χειροπιαστά αποδεικτικά στοιχεία. Ευχαριστούμε η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Δεν ε, με ενδιαφέρουν τόσο η ακρίβεια των στοιχείων, διότι όταν υπήρχε ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, ε, ακόμα και αν δεν είναι υψηλά τα υψηλοί δείκτες, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Γι' αυτό λοιπόν ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευαισθησία στον θόρυβο, ναι, επειδή ζούμε σε ήρεμε σε ήρεμε περιοχές, σε ήρεμου χώρους. Αυτό το ξεχνάμε συχνά. Συχνά όμω οι αρχέ δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή του για να περιορίσουν το φαινόμενο. Από ιατρική σκοπιά όλοι κατέδειξαν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Δηλαδή υπάρχουν θόρυβοι που προκαλούν ε, προβλήματα καρδιο καρδιολογικές ε, παθήσεις, ε, ακόμα και δυσκολίες μάθησης από πλευρά των παιδιών. Κανένα οψία μου λοιπόν θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 7, όπου αναφέρεται πως ε, μόνο κατά από ορισμένες συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση μιας χαρτογράφησης ακουστικής στρατηγικής φύσης. Δηλαδή μόνο όταν υπάρχει πάνω από κάποιος αριθμός αυτοκινήτων, σιδεδρόμων κλπ τα οποία κυκλοφορούν. Αυτή λοιπόν η υποχρέωση θα πρέπει να υφίσταται για όλες τις ε, περιοχές, για όλες τις επικράτειες και να μετράται η έκθεση στον, ε, στην υγορύπανση και να υπάρχουν τα πρόγραμματα δράσης για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η οδηγία είναι σωστή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Έχω μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία ακούσαμε από τους ε, αγορητές. Ε, για το γεγονός ότι τα στοιχεία τα οποία ε, έχουν συλλεγεί. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι δεν είναι αξιόπιστα και δεν ε, βεβαιώνουν τις επιπτώσει του χορύπανση στην ανθρώπινη υγεία. Όπως ε, μας ενημερώσατε λοιπόν όλοι σας, θα ήθελα να μάθω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε ανάλυση του θέματος και αν έχει προβλέψει συγκεκριμένες δράσεις και, ποιε, και τι επιπτώσεις θα έχουν οι δράσεις αυτές στην οικονομία των μελών, στην μεταφορά των ε, εμπορευμάτων κλπ. Ειδικά θα μιλάω για τα νέα κράτη-μέλη, δηλαδή ε, τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Γνωρίζετε ότι αυτή η τόσο δογματική θέση σύμφωνα με την οποία πρέπει να καταργήσουμε, να απαλείψουμε τον θόρυβο, δίχως ε, να νοιαστούμε για τις οικονομικές συνέπειες ε, που θα προκαλέσει κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου και στη δική μου τη χώρα ε, είναι δύσκολο να γίνει δεκτό. Εν ολίγης, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις δράσεις που θα προτείνετε και θα αναλάβετε και που αφορούν το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα να εξετάσετε επίσης και τις γνώμες των ε, μεταφορών, των μεταφορέων συγγνώμη, των κρατών, κρατών όπως η Πολωνία όπου η συγκεκριμένη βιομηχανία μπορεί να υποστεί τεράστιες ζημιές σε ό,τι αφορά την λειτουργία, τι δραστηριότητε τη, αλλά και την απασχόληση. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θα ήθελα να επαναλάβω αυτή την ερώτηση. Έχετε δείκτες, έχετε υπολογίσει, έχετε αναλύσει. Πώς αυτές οι απόψεις ε, θα επηρεάσουν αρνητικά τους, ε, την ανταγωνιστικότητα των, ε, των εταιριών αυτού του αυτοκινητικού κλάδου. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μερικέ ερωτήσει. Για να δουλέψει καλά πρέπει να κοιμάσαι καλά. Γιατί άμα κοιμάσαι άσχημα δεν δουλεύει καλά. Εμεί περιμένουμε όλοι να αποδίδουν και αν δεν μπορεί κάποιο να κοιμηθεί καλά θα πρέπει να προγραμματιστούμε τι θα γίνει. Πέρα από τον αριθμό των νεκρών, αλλά ότι ο θόρυβο βλάπτει την υγεία είναι σαφές ή την επηρεάζει. Ίσως ακούσουμε και περισσότερα. Ακούσαμε επίσης ότι εδώ και χρόνια, ενώ όχι δεκαετίε, η την επηρεαζει σω ακουσουμε και περισσοτερα ακουσαμε επιση οτι εδω και χρονια αν οχι δεκαετιε η ευρωπαικη επιτροπη ε, ασχολείται με το θόρυβο, με τις οδηγίες, αλλά για τις εκπομπές έχουμε οριακές τιμές για τις πόλεις και για τους δρόμους. Ε, ε, ε, για, για τα χιλιόμετρα ας πούμε, αλλά για το θόρυβο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πότε θα έχουμε και οριακές τιμές για το θόρυβο, ανεξαρτήτως από τις βλάβες στην υγεία τους νεκρούς. Υπάρχει βλάβη, βλαβερή επίδραση στην υγεία που θα πρέπει να μειωθεί. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Ερώτηση δεύτερη. Νομίζω πριν από 30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εξαγγείλει ότι θέλει να βάλει ε, ως κανόνα ταχύτητα στην πόλη τα 30 χιλιόμετρα. Ε, μόνο το 10% των πιο ευάλωτων χρηστών του δρόμου, ποδηλάτες ε, ε, και πεζοί και τα λοιπά, παθαίνουν σοβαρό δυστύχημα όταν είναι 30 χιλιόμετρα κυκλοφορία, ενώ όταν είναι 50 το 80% για το θόρυβο θα πρέπει να ισχύουν αντίστοιχα. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να είναι στάνταρη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα και θα μειωθεί και ο θόρυβο. Πότε θα μας φέρετε τέτοια πρόταση. Και τρίτον, έχω την εξή ε, εμπειρία. Σε θορυβώδεις περιφέρειες ε, δεν ζουν εκείνοι που είναι πιο εύποροι και πιο λεφτάδες. Ε, κοντά σε αεροδρόμια δεν ζουν άνθρωποι που κερδίζουν 5.000 ευρώ το μήνα. Έχει πουλήσει το σπίτι του εδώ και καιρό το οποίο θα υποβαθμίζεται και θα χάνει την αξία του. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο κοινωνική διάσταση. Ποιε είναι εκείνε οι κοινωνικέ ομάδε, οι ομάδε του πληθυσμού που πλήττονται και πώ σκοπεύετε να το λύσετε. Εδώ τελειώσαν οι ερωτήσει. Έχετε πέντε λεπτά έκαστο για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Thank you. Thank you very much. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη μητρική σα. Ναι, αλλά δεν ξέρω την ορολογία. <laughs> I admit this. Ομολογώ ότι τα ξέρω καλύτερα στα αγγλικά παρά στα γερμανικά. Ήταν πολλές ερωτήσεις και δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ήταν χρήσιμο για μένα να το ακούσω. Μέσα μόνο, σε μόνο πέντε λεπτά πρέπει να επικεντρωθούν σε κάποια βασικά σημεία. Πολλές ερωτήσεις είχαν να κάνουν με τους πρώιμους θανάτους και τους αριθμούς που ανέφερα. Με τους πρόωρους θανάτους. Αυτό δεν είναι κάτι που το επινοήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι από την έκθεση της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Ε, είναι αριθμός από το 2014 και βασίστηκε σε άλλες μελέτες και αυτοί οι αριθμοί μάλλον είναι και χαμηλότερη από την πραγματικότητα. Εξ όσων γνωρίζω έχουν υπολογιστεί, γιατί δεν τους έχω υπολογίσει μόνος μου, βάσει των επιδημιολογικών μελετών που δείχνουν τη σχέση μεταξύ θορύβου και αυτό που ονομάζεται τα ε, ανόφλια υγείας. Δηλαδή ε, διαταραχές του ύπνου, καρδιοαγγειακές παθήσεις και άλλες ψυχολογικές διαταραχές. Αυτές είναι οι βασικές επιπτώσεις του θορύβου. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες σχετικά και αποδεικτικά στοιχεία και δείχνουν ότι υπάρχει συσχετισμός. Ο ΠΟΕ, ο μάλλον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εργάζεται για τα θέματα αυτά με τη συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμόνων και προσπαθεί να καθορίσει τον σαφή ε, συσχετισμό μεταξύ της έκθεσης στο θόρυβο και των επιπτώσεων στην υγεία. 30-40.000 ε, πρόοροι θάνατοι της ΥΟΣ, αναλόγως με το πόσοι είναι εκτεθειμένοι σε τι επίπεδα θορύβου και μετά με βάση αυτή τη σχέση μπορεί κανείς να υπολογίζει τις άμεσες συνέπειες. Εάν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα σας έλεγα να διαβάσετε την έκθεση «Θόρυβο στην Ευρώπη 2014», μελέτη στην οποία βασιστήκαμε κι εμείς και κυρίως και τις κατευθυντήριες γραμμές για το θόρυβο, που αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται σε φάση αναδιατύπωσης, θα τα βρείτε σύντομα στο ίντερνετ αφού ε, επικαιροποιηθούν. Ως προς τους ε, αριθμούς, λοιπόν, από εκεί ήταν η παραπομπή. Επίσης, τέθηκαν και άλλες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω μία-μία. Σε ό,τι αφορά το θόρυβο από τους σιδηροδρόμους, τα βαγόνια, τις ράγες, αυτό δεν είναι, είναι μέσα στο πεδίο της Γενικής Διεύθυνσης από την οποία προέρχομαι και στην οποία εργάζομαι. Εμείς κοιτάζουμε πώς να βελτιώσουμε τα πράγματα σε σχέση με την υποχωρήπαρξη. Η οδηγία για την οποία συζητάμε είναι οδηγία πλαίσιο περισσότερο. Υπάρχει πάντως σχετικό πρόγραμμα και τα σχετικά κονδυλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αν μπορούμε να έχουμε ένα ειδικό κονδύλι, ένα ποσό για να αποσύρουμε τα παλιά βαγόνια, τις παλιές αμαξοστοιχίες όπως είπε ένας ε, Γερμανός βουλευτής, θα μπορούσα να το αναφέρω αυτό στην υπηρεσία μου, δεν το έχουμε σκεφτεί από μόνοι μας, αλλά να το πω στους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης μου. Δεν ξέρω πόσο χρόνο πραγματικά θα μου δώσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις λεπτομερώς. Ένα στοιχείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι μάλλον το γιατί δεν έχουν γίνει περισσότερα έχει να κάνει με πολλά άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί. Εδώ είμαι υπάλληλο τη Επιτροπή. Δεν είμαι επιστήμονας πρέπει στην πράξη με αυτά και δεν μπορώ να ε, αποφασίσω τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Ούτε πολιτικός είμαι. Ε, δεν γνωρίζω το κόστος, ούτε τι οικονομικέ διαστάσεις του θέματος. Είναι ένα αριθμό μόνο θα σα αναφέρω, διότι η μελέτη που εκπονήσαμε πριν από λίγο καιρό ε, λέει μιλάει για 40 δις ετησίως κοινωνικό κόστος από το επιπτώσεις του θορύβου. Αυτό έχει να κάνει με το σύστημα υγείας, την επιβάρυνσή του δηλαδή, με τις απώλειες ζώων, με τις δυσκολίες στην στέγαση. Γιατί δεν έχουν γίνει λοιπόν περισσότερα διότι η οδηγία για το θόρυβο λειτουργεί, ε, έχει εγκριθεί μάλλον το, έχει τεθεί σε ίσχυ από το 2002. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα αξιολογούμε το τι συμβαίνει βάσει αυτή τη αξιολόγηση και αν μα οδηγήσει συλλογικά συμπεράσματα ε, η μελέτη μα θα μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώ πρέπει να γίνει με το θόρυβο για να σα πούμε και τα αποτελέσματα σε σχέση με τα όρια, τα επίπεδα θορύβου. Σε κάθε περίπτωση πάντω θα δούμε όλε τι διαφορετικέ επιλογέ που υπάρχουν και θα κάνουμε τη σχετική πρόταση. Αυτή ήταν η βασική μα ιδέα. Να δω αν ξέχασα κάτι σημαντικό, επιπτώσει στον ανταγωνισμό. Ναι, σαφέ. 40 δι ετησίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κόστο θορύβου, πανάκριβο. Όρια ταχύτητα από την οδηγία για το θόρυβο. Δεν νομίζω να επηρεάζεται την οδηγία για το θόρυβο, αλλά τα κράτη-μέλη αν θέλουν από μόνα τους μπορούν ε, κατόπιν να ορίσουν ε, όρια δικά τους για να αναχαιτήσουν τα προβλήματα του θορύβου. Είναι ο φθηνότερο τρόπος τα όρια ταχύτητας. Μπορεί να περιορίσει και τα ατυχήματα μάλιστα. Αλλά αυτό είναι θέμα εξισορρόπηση στα κράτη-μέλη, στι περιοχέ, στι επιμέρου τη και ούτω καθεξής. Είναι ένα σημείο ισορροπίας που ακόμη δεν έχει βρεθεί. Ελπίζω ότι τα κάλυψα όλα στον τόσο λίγο χρόνο που είχα. Α, ναι, η κοινωνική διάσταση. Καλώς και μου το θυμίζετε, διότι έχουμε πονήσει δύο μελέτες, σας τις συστήνω Αναπιφύλακτα. Ο, ε, η μία ονομάζεται θόρυβος και επιπτώσεις στην υγεία, Εάν δεν μπορείτε να τη βρείτε, απευθυνθείτε απευθεία σε εμά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Από την Υπηρεσία για την Σχετική Πολιτική. Η μία ονομάζεται Επιπτώσει του θορύβου στην υγεία και η άλλη ακριβώ αυτό που ρωτήσατε, κοινωνική διάσταση στην υγεία. Δεν έχω χρόνο να σα εξηγήσω. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι υπάρχει πολύ περίπλοκο σχετισμό μεταξύ θορύβου και υγεία διότι δεν ζουν τις θορύβοδε περιοχέ οι περισσότεροι και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν και τι αρνητικέ συνέπειε. Αλλά είναι και δύσκολο να κανεί κανείς ε, τι αρνητικέ κοινωνικέ συνθήκε από τι επιπτώσει του θορύβου του ίδιου, της ίδιας. Υπάρχουν λοιπόν και κοινωνικέ και οικονομικέ συνέπειε από το θόρυβο. Μπορείτε να βρείτε τι σχετικέ μελέτε στο διαδίκτυο και πραγματικά συνοψίζουν τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εσείς έχετε το λόγο κύριε Γότη. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ για κάποιες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολήθηκε και ο κύριος Μπέργερ. Θα φροντίσω να αντιμετωπίζω μια και δύο από αυτές. Δεν έχω χρόνο να σας ε, παρουσιάσω τα υπόλοιπα slides, τις διαφάνειες. Ο κ. Μπέργκεν αναφέρθηκε ότι υπάρχουν κάποιες ε, οριακές τιμές στην ε, σχετική οδηγία περί χορύπανσης. Θα υπάρχουν λόγια τους οποίους χρειάζεται να υπάρξουν αυτές οι οριακές τιμές και η αντιμετώπιση των συγχωρήπανσης ε, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο. Η σχετική οδηγία περί χορύπανσης και πηγών θα πρέπει να εφαρμοστεί για κάποιες, κάποιους τρόπους μεταφοράς παραδείγματος χάρη που έχουμε στον συνδρομικό τομέα όπου έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος το ζήτημα των ελαστικών έχει μειώσει την ηχορύπανση που προκαλείται από τα λάστιχα. Η πρόοδος που έχει επιτύχει και η βιομηχανία σε διάφορους κλάδους είναι αποτελεσματική και έχουν φροντίσει να μειώσουν επίσης τον ήχο οι εταιρείε ε, αεροναυπηγικής το θόρυβο με οποίο εκπέμπουν τα αεροσκάφη. Οι διάφοροι τρόποι μεταφορών επηρεάζουν διαφορετικά τους ανθρώπους. Χρειάζονται λοιπόν αυτά, αυτές οι στη τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Και επηρεάζουν αμφίβολα και την οικονομική δραστηριότητα εάν επιτευχθεί η ανταρμόνιση. Υπάρχει λοιπόν και δυνατότητα να μην περαστούν ε, υποχρεωτικέ όλες αυτές οι ε, οδηγίε. Ο κύριος Μπέργκερ πάλι. Ναι, μια ερώτηση που Η μέρα του θορύβου, ε, κάποια στιγμή τον Απρίλιο είναι, στις 27. Κάθε χρόνο υπάρχει μέρα κατά του θορύβου, τον Απρίλιο, τόσο του μήνα. Ευχαριστώ πολύ vielen Dank Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Μάθαμε και κάτι. Πάει λοιπόν το πρώτο πάνελ. Ευχαριστώ ε, όλους τους ομιλητές, όλους ε, τους βουλευτές που έκαναν ερωτήσεις και πάμε μέσα στο επόμενο πάνελ. Σας παρακαλώ να κατεβείτε για να έρθουν οι επόμενοι. Und Herr Wolfgang Eberle, Markus Hecht. Wolfgang Eberle, Markus Hecht, και Wiltord Groll. Παρακαλώ, ελάτε.

με στο επόμενο πάνελ ε, για το θόρυβο στις ε, ε, αυτοκινητοδρόμους, στους σιδηροδρόμους και ε, στις αναέριες μεταφορές. Ο Wolfgang Έμπερλε έχει πρώτο το λόγο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας Τροφίμων και Δασών του κρατηδίου της Ρινανίας Παλατινάτου. Έχετε το λόγο κύριε Έμπερλε. Ebenfalls 10 minuten. Για δέκα λεπτάκια εσείς. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω το θέμα μας από τη Ρινανία Παλατινάτο, ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο της Γερμανίας, αλλά και γενικότερα από τη Γερμανική Εταιρεία Ακουστικής. Ε, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αξιολογείται σε πολύ ψηλό επίπεδο και είναι αντικείμενο αλλά και στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό ισχύει και για την προστασία από το θόρυβο, ιδιαίτερα από το θόρυβο στην κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους. από 55 δεσιμπέλ και πάνω, 24 ώρες το 24ωρο, ο θόρυβος ενοχλεί ή επηρεάζει σοβαρά την υγεία. Γύρω από τα μεγάλα αεροδρόμια ζουν λιγότεροι πολίτες μεν, αλλά ε, ενοχλεί πολύ περισσότερο θόρυβο στο αεροπλάνο από ότι του σιδηροδρόμου ή του αυτοκινητοδρόμου. Αυτό το έχει δείξει μια μελέτη που μελέτησε τέσσερα μέσα μεταφοράς. Στο σιδηρόδρομο αυτό που έχει σημασία είναι η νυχτερινή κυκλοφορία, εμπορευματικέ μεταφορές ε, πάνω στις ράγες. αλλά αυτό αφορά λιγότερους ανθρώπους γιατί είναι περιορισμένες οι διαδρομές που μελετησε τεσσερα μεσα μεταφορας στο σιδηροδρομο αυτο που εχει σημασια ειναι η νυχτερινη κυκλοφορια εμπορευματικε μεταφορες πανω στι ραγες αλλα αυτο αφορα λιγοτερους ανθρωπους γιατι ειναι περιορισμενες οι διαδρομες που κανουν ε, τα εμπορεύματα αυτά. Κάθε χώρα και κάθε κράτος συνδέεται με ένα οδικό δίκτυο και ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και καλά κάνει. Αλλά ε, αυτό σημαίνει ότι είναι πανταχού παρόν ο θόρυβος 74 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι, μάλιστα 200.000, ε, επηρεάζονται από το, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ και ε, μια αρμόδια γερμανική υπηρεσία το 2008 και το 2009 έχουν δημοσιεύσει στοιχεία για τη Γερμανία για τα παιδιά. Όσο περισσότερη έκθεση έχουν σε θόρυβο, ε, τόσο των παιδιών, τόσο χαμηλότερη είναι η κοινωνική κατάσταση. 12,8% ε, ε, είναι τα παιδιά μεσοαστικά υψηλά κοινωνικά ε, στρώματα, ενώ 27,8 το υπερδιπλάσιο είναι από κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Δεν υπάρχει ε, όμως ε, πανάκια που να επιτρέπει να μειωθεί κατά 10% και παραπάνω ε, ο θόρυβος ή κατά 5 δεσιμπέλ. Ε, υπάρχει τρόπος με τεχνικές, με συγκεκριμένες ασφάλτους ή συγκεκριμένες ράγες να μειωθεί ε, η έκθεση στο θόρυβο, η παραγωγή θορύβου κατά 5-10 δισιμπέλ. Στον αυτοκινητόδρομο αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Σε πολλές ε, περιπτώσεις και με πολλούς τρόπους ε, ο θόρυβος επηρεάζει. Επηρεάζει την επικοινωνία, την ποιότητα ζωής, ενοχλεί τον ύπνο και υπάρχει κίνδυνος εγκεφαλικό και καρδιακή προσβολή. Αυτό φάνηκε από τη μελέτη Νόρα. Υπάρχει σύνδεση ε, μεταξύ του θορύβου από την κυκλοφορία και την εμφάνιση κατάθλιψης. Αυτό πραγματικά μας εξέπληξε. Από ό,τι φαίνεται ε, υπάρχουν κάποιες δόσεις που ε, προκαλούν συγκεκριμένες βλάβες για την υγεία. Βλέπετε εδώ τους άξονες χ και ψ, κάθετο και οριζόντιο για την προστασία από θόρυβο στην Ευρώπη είναι σημαντικό βήμα. Τέτοια αποτελέσματα ερευνών να αξιολογούνται, να μελετώνται και να ε, μεταφράζονται οι δόσεις. Αυτό γίνεται αυτό τον καιρό με την επικυροποίηση ε, του παραρτήματος της οδηγίας αυτής. Φτάνει όμως αυτό το βήμα. Ε, είναι ο θόρυβος Βραβερό για την υγεία, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το κατόφλι. Δεν υπάρχουν κατώτατες τιμές. Ε, και ε, είναι ένα ε, ύπουλος εχθρός. 9% ε, κίνδυνο για κατάθλιψη, τι σημαίνει. είναι αμεληταία ποσότητα, είναι παράπλευρη απώλεια, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ανεχθούμε ή όχι. Ε, αυτά θα πρέπει να αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό ή σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο από τον νομοθέτη. Δεν μπορεί να το απαντά ο κάθε Δήμος, ε, διότι συνδέεται με αυτό ε, ο υποχρεωτικός ή μη χαρακτήρας, άρα και η απαραίτητη χρηματοδότηση. Ως προστασία λοιπόν από το θόρυβο υπάρχουν διάφορα μέτρα, τα οποία τα γνωρίζετε θα ήθελα να σας μιλήσω εδώ ε, στην καταπολέμηση του θορεύου στην πηγή, σε πιο αθόρυβους τρόπους και βεβαίως υπάρχουν και κάποια ε, παράθυρα που μπορεί κάποιος να βάλει στο σπίτι του διπλά τζάμια και τριπλά αν δεν ε, υπάρξει ε, άλλη δυνατότητα καταπολέμησης. Ε, συνδυασμός μέτρων είναι αυτός ε, που βοηθάει. Ε, σε ό,τι αφορά στη Γερμανία, από το 2000, μάλλον από το 1992 έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα γιατί δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Ε, με τη Συμφωνία του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την απέτηση να αυξηθεί η ποιότητα του αέρα, να βελτιωθεί μάλλον, ε, φαίνεται ε, ότι στο επόμενο μέλλον, στις επόμενες δεκαετίες θα αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορούμε στις πόλεις. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί ό,τι είναι καλό για το περιβάλλον και την ατμοσφαίρα είναι καλό και για την καταπολέμηση του θορύβου. Για να ε, έχουμε συγκεκριμένους στόχους χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι για να μπορέσουν να τηρηθούν. Μέτρα λοιπόν κατά πολέμηση του θορύβου στη πηγή ε, για να πληρώνει ακριβώς ο ρηπαίνων. Στην Ευρώπη έχουμε ένα κανονισμό τη 16 Απριλίου 2014 ε, για ε, το θόρυβο που εκπέμπουν τα φορτηγά. Η οδηγία του 2014 είχε μια ευκαιρία αλλά χάθηκε. Το 2037 προβλέπεται να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη και να μειωθεί ο θόρυβος κατά έναντι δισιμπέλ μόνο. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2021 όμως υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να κάνει μια μελέτη και να τη δημοσιεύσει. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης μπορεί να κάνει πρόταση νομοθετική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό ε, μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένη οδηγίας. Άλλες δυνατότητες ε, έχουν τα ελαστικά ε, των ε, αυτοκινήτων ή σε κάποιο ειδικό υλικό με το οποίο καλύπτονται οι ράγες, οι τυροτροχές. Ή το οδόστρωμα. Ο θόρυβος αφορά πολλούς κλάδους και πολλά επίπεδα αρμοδιότητας. Άρα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολλές οι γενικές διευθύνσεις. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια συνεκτική πολιτική και υπάρχει η πράσινη βίβλος του 1996 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει πλέον λευκή βίβλος για τη μελλοντική πολιτική. Είναι σημαντική η στόχη, είναι πολύ φιλόδοξη και σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν υπάρχει απέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανευρωπαϊκή, για την καταπολέμηση του θορύβου στην πηγή με δεσμευτικούς στόχους και, και με φιλόδοξους. Συνοψίζω. Σήμερα οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες, αλλά έχουν πολλά εμπόδια να αντιμετωπίσουν και η βασική δυσκολία κατά την άποψή μου είναι η εξής είναι πολύ λίγα τα μέτρα πολέμηση του θορύβου που μπορούν ουσιαστικά να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Θα πρέπει να προστατεύεται σε υψηλό επίπεδο η δημόσια υγεία. Στον αυτοκινητόδρομο δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Για να προστατευθούν λοιπόν ε, οι ομάδες του πληθυσμού που έτσι κι αλλιώς και με βάση την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής ε, χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης, ένα οδικός χάρτης για μια συνεπή ευρωπαϊκή πολιτική. Αφετηρία θα πρέπει να αποτελέσει η μετεξέλιξη ε, της Πράσινης Βίβλου του 1996 σε μια λευκή βίβλο για την πολιτική. Αρχής γενομένης λοιπόν από την Πράσινη Βίβλο ε, η οδηγία έθεσε το απαραίτητο πλαίσιο. Ξέρουμε πολύ ε, ξεκάθαρα σήμερα ποιο είναι ο θόρυβο στην Ευρώπη και πώ είναι οι πολίτε που πλήττονται. Αλλά μα λείπει το δεύτερο βήμα. Τώρα, ποια μέτρα είναι αυτά που θα εφαρμοστούν έτσι ώστε να ε, μεταξελιχθεί η συγκεκριμένη οδηγία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ελάχιστε ε, προποθέσει για την προστασία τη δημόσια υγεία με συγκεκριμένου στόχου. Ενιαίου στόχου πρέπει να έχει η Ευρώπη Ε, υπάρχει ε, σύμφωνη ρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που προβλέπει τα 55 δεσιμπέλ. Ε, έστω και τα 65, αν είναι το ανοιχτό όριο. Κατά την άποψή μου θα ήταν αυτό κάτι που θα μπορούσε να συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη-μέλη να βάζουν στόχους προστασίας στα πλαίσια του τεχνικά εφικτού και στα πλαίσια των κατόπους δυνατοτήτων με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Για μια βιώσιμη κινητικότητα θα πρέπει η οδηγία καταπολέμησης του θορύβου να γίνει οδηγία πλαίσιο ε, και να συμπεριλαμβάνει και ρυθμίσεις για τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητή, ο καθηγητή Χέκτ από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο δηλαδή, του Βερολίνου. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε σήμερα για να σας ε, κάνω αυτή την παρουσίαση μέσω των διαφανειών σημαντική, ε, μετριασμός της, ε, του δωρίου μπορεί να προκύψει από την σχετική οδηγία και από την ε, οδηγία TSI. Ε, τώρα το πώς θα μειωθεί ο, ο θα σας το εξηγήσω με την επόμενη διαφάνεια. Θα πρέπει να δίνουμε αυτή την ανάγνωση στην ε, διαφάνεια. Εδώ υπάρχει η περιοχή του, μια πόλη στο Ρήνο, όπου ο θόρυβος είναι ψηλός. Πάνω από 55 decibel, είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε επανειλημμένα. Νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή, θα πρέπει να διατηρηθεί στην Γερμανία. Περισσότερο από 6 εκατομμύρια άνθρωποι γνωρίζουν επίπεδα της τάξης του 85, δεσιμπέλ. Πραγματικά απίστευτο. Έχετε λοιπόν εδώ πολύ συχνές διαμαρτυρίες κατά αυτής της κατάστασης, της συγχωρήπανσης. Τι γίνεται. Εδώ πρόκειται για κάποια εθελούσια μέτρα τα οποία υπάρχουν δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες διότι ο χρόνος πιέζει. Απλά θα σας δώσω μια ιδέα σχετικά με τι κάνουν οι σχετικές αρχές οι οποίες έχουν υποβάλει κάποια ερωτηματολόγια όπου ρωτούν αν είστε, και κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα μετριασμού και βλέπετε ότι 1% μόνο είναι ικανοποιημένο και το 99% δεν είναι ικανοποιημένο. Τι συμβαίνει, ε, Τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την ε, επίτευξη του στόχου των 55 δεσιμπέλ είναι ο μητριασμός ε, του θορύβου στην πηγή. Και τι έχει γίνει από το 2003 για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο ε, του θορύβου θα πρέπει να γίνεται λοιπόν στην πηγή και το μόνο κράτος που το ε, εφάρμοσε ήταν η Ελβετία. Καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το πέτυχε. Η μείωση της συγχωρήπανσης ε, θα πρέπει να γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων, των σειρμών, των σιδηροτροφιών και να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία εφάρμοσε και η Ελβετία μέχρι τώρα. Το βελτίωση της... Ε, η εφαρμογή μάλλον της οδηγίας θα πρέπει να βασίζεται δύο στοιχεία. Η διαχείριση του ήχου, η διαχείριση του ήχου θα πρέπει να στοχεύσει στην επίτευξη του στόχου του 55% και να μην ε, συνεχιστεί η κατάσταση που ε, ισχύει μέχρι τώρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν κατά μήκο των σύντογραμμών ε, κέντρα ελέγχου για την μέτρηση των, ε, της συγχωρήπανσης παραδείγματα στην Ελβετία από το 2003 έχουμε αυτά, στις, ε, αυτά τα κέντρα ελέγχου του συγχωρήπανσης Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή η παρακολούθηση τους, χορύπανση κατά μήκος των σιδηροτροχιών. Κάτι επίση το θέμα είναι το, αφορά τον, τον έλεγχο του θόρυβου από TSI. Τις πιο πολλές φορές έχουμε προβλήματα από το, από το σύστημα της των, των τρένων. Σήμερα, εάν υπάρχει πρόβλημα, να ε, σας πω ένα, παρα... ένα ένα παράδειγμα. Η εταιρεία Bombardier έκλεισε την, ε, το τμήμα της για τον έλεγχο των, ε, της ηχορύπανσης for the competitiveness of our products. Και Φυσικά όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Διότι αυξάνει το κόστος. η, ποιότητα των, των διότι τον θόρυβο δεν τον προκαλούν μόνο η τροχή, αλλά προκαλείται και από τις τροχές. Να σας πω τώρα ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές λύσεις. Ήδη από το 1996 έγιναν κάποιες δοκιμές στην Βαβαρία και κατέδειξαν ότι ήταν δυνατόν να επιτευχθούν λιγότερα κατα, ε, λιγότερο από 25 δεσιμπέλ στην ε, Ιαπωνία έγιναν αυτές οι δοκιμές με το τρένο ταχύτητα του 300 χιλιόμετρων την ώρα με μείωση παράλληλα 20 δεσιμπέλ του ήχου που εκπέμπουν έχουμε και την περίπτωση των ε, ε σειρμών που ε, προκαλούν 12% η χορύπανση Τώρα, για ποιο λόγο οι κανονισμοί της Ένωσης έχουν τις απαιτήσει Euro 4, Euro 5 και αν κοιτάξετε τα όρια που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ε, εάν υπήρχε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομίζω ότι και οι Αμερικανοί θα ακολουθούσαν μια παρόμοια νομοθεσία. Αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό, ζήτημα κλειδί. Ο θόρυβος από TSI Ευχαριστώ πολύ. Ο Βίτολτ Γκρόλ ακολουθεί από τη Βαρσοβία για, ε, στο Αρμόδιο Σιδηροδρομικό Ινστιτούτο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην σύντομη παρέμβασή μου θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα πρόβλημα και να σας πω τι γίνεται με το πρόβλημα του θορύβου από τους στην Πολωνία συγκεκριμένα. Ο μέσος κάτοικος είναι εκτεθειμένο σε διαφορετικές πηγές θορύβου των σιδηροδρομικών, των αεροπορικών μεταφορών, των οδικών και των βιομηχανικών μονάδων. σε γενικές γραμμές ε, οι πηγές αυτές του ρήπου βρίσκονται παντού γύρω από τους μέσους κατοίκους αλλά από μια μελέτη προκύπτει ότι το ποσοστό των ατόμων που θεωρούν ως πηγή ενόχλησης τον θόρυβο είναι χαμηλότερο στην περίπτωση των σιδηροδρόμων και πιο υψηλό σε περιπτώσεις άλλων ειδών μεταφοράς. Αυτό δείχνει ότι είναι διαφορετικό το μερίδιο του πληθυσμού που είναι κεθυμένο στο θόρυβο. Κατ' εμέ, οι συστάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία θα πρέπει να ορίζουν σε ανώτερο επίπεδο τα 55 δεσιμπέλ για τον θόρυβο στην πηγή και τις διάφορες δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο. Όλες οι πηγές θορύβου προκύπτουν από κάποιο είδος μεταφορά συνήθως. Το να προβλέψουμε ένα όριο που ε, πλήττει την ανταγωνιστικότητα ενός είδους μεταφοράς σε σχέση με ένα άλλο είδος, δημιουργεί τελικά έναν επιθύμητο, ένα αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Και τελικά μπορεί κανείς να είναι και περισσότερο εκτεθειμένο στο θόρυβο αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έκθεσης. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, η μάχη κατά του θορύβου είναι ένας αγώνας για τον περιορισμό του θορύβου στις πηγές. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι, άλλες μέθοδοι. Το γεγονός, οι προσπάθειες ε, περιορισμού του θορύβου εξαρτώνται από τον πληθυσμό, τις οδικές υποδομές, την ταχύτητα, το είδος του υλικού που κυκλοφορεί ε, στις διάφορους, στους διάφορους δρόμους και ούτω καθεξής. Οι διάφοροι παράγοντες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο ποσοστό των ατόμων που πλήττονται από προβλήματα χορύπανσης. ασχέτως της καταπολέμησης του θορύβου στην πηγή. Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων Μεταξύ των, αυτο, ε, παραστάσεων που είδαμε στις προηγούμενες διαφάνειες βλέπετε την ε, πυκνότητα του πληθυσμού εδώ στην ε, Ευρώπη. Στην Πολωνία είναι σχετικά αραιή η κατοίκηση της χώρας σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία, οι κάτω χώρες ή η Ελβετία. Ο θόρυβος από τους σιδηροδρόμους προκαλείται από διαφορετικούς παράγοντες. Όλοι αλληλοσχετίζονται και επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα την κατάσταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Πολωνίας. Στην Πολωνία αναλύσαμε περίπου χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, εδάφους που διασχίζουν οι σιδηρόδρομοι. Βλέπετε τις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα στο χάρτη. Στα νότια της χώρας οι περιοχές αυτές αφορούν και αστικά κέντρα. Κάναμε ανάλυση για τον πληθυσμό των αστικών κέντρων και στην Πολωνία το ποσοστό του πληθυσμού ε, που είναι εκτεθειμένο στον θόρυβο είναι χαμηλότερο. Είναι σχετικά χαμηλό μάλλον. 2% στην έκθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας και 0,5% στην ε, διάρκεια της νύχτας. Στην Πολωνία υπάρχουν κάποιες δράσεις για την αναχέτηση της ηχορύπανσης λόγου χάρη στην, ε, ε, στον εξοπλισμό των ε, αμαξοστοιχειών με σύνθετα υλικά για την πέδηση. Εδώ αυτά εξαρτώνται από την αξία και από την ποιότητα του υλικού, από τον τρόπο που φρενάρουν τα τρένα. Όσο πιο συχνά φρενάρουν οι σειρμοί, η διαφορά μεταξύ του θορύβου που προξενείται τα σύνθετα υλικά και τα κλασικά συστήματα πέδησης είναι πολύ μεγαλύτερη. Ως προς το θόρυβο ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η συντήρηση των ε, βαγονιών των ίδιων, των σειρμών. Ιδίως όταν δεν υπάρχουν εργαλεία για να παρακολουθήσουμε, να ελέγξουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα βαγόνια. Οι πληροφορίες αυτές ε, σε σχέση με την Πολωνία μας, μας φέρνουν στις εξής ερωτήσεις στους εξής προβληματισμούς. Σε γενικές γραμμές, ο θόρυβος που προκαλείται από τους υδροδρόμους είναι κίνδυνος ε, κατά της υγείας των Πολωνών πολιτών. Όπως επιβεβαιώνει η έκθεση του Γενικού, ε, της Γενικής Διεύθυνσης για την παρακολούθηση των σιδηροδρόμων, δεν είναι η βασική πηγή προβλημάτων από την ηχορύπανση σιδηρόδρομων στην Πολωνία. Περισσότερο πρόβλημα προκαλούν οι οδικέ μεταφορέ. Εδώ έχουν ε, να κάνουν πολλοί άλλοι παράγοντε, όπω η πυκνότητα του πληθυσμού λόγω χάρη. Στην Πολωνία είναι σχετικά χαμηλή. Ή η, η ταχυτητα Υπάρχει ίσω καλύτερη οργάνωση στου σιδηροδρόμου, και επίσης το γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοι δεν αφορούν τόσο πολύ τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα, στην αγορά της Πολωνίας, στην Πολωνία υπάρχουν πάνω από 200, 200 φορείς εμπορευόμενοι βαγονιών, αλλά μόνο 108,5 ε, αμαξοστοιχειών, ε, μικρό ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά το 85% είναι εμπορικά, ε, εμπορική σειρμή, ενώ το 15% μόνο είναι το υπόλοι, οι υπόλοιπες κατηγορίες σειρμών. Εδώ έχουμε ένα στόλο από βαγόνια εμπορεύματα μεταφορών που είναι συγχρονισμένα με τις απαιτήσει TSI Noise για τον θόρυβο. Έχουμε περίπου δηλαδή 2.000 ε, περίπου 400 βαγόνια που είναι σε αυτή τη ε, φάση. Κάποια όμως ε, βαγόνια έχουν ε, τροχούς ε, ενιαίους χωρίς ελαστικά. Τα 17.000 περίπου, ενώ τα 60.000 το αντίθετο. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν των, εμπορευματο... των εμπορευματικών ε, σειρμών χωρίς ελαστικά βρίσκεται στην Πολωνία. Εάν θέλαμε να τα ε, εφαρμόσουμε αυτά σε παλιές αμαξιοτεστοιχίες για να φτάσουν στις προδιαγραφές ε, TSI για το θόρυβο, τι θα συνέβαινε. Πρώτα απ' όλα θα ήταν πολύ μεγάλο το κόστος. Μπορεί επίσης να επλείται εδώ η ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά. Ο κίνδυνος είναι η αγορά να κατακλειστεί από τις οδικές μεταφορές στην ουσία. το κόστος που θα προέκυπτε από την προσαρμογή στις προδιαγραφές TSI στην Πολωνία θα έφτανε περίπου το μισό δις ευρώ και αυτό επειδή στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνταν σύνθετα υλικά για τα συστήματα πέδησης θα έπρεπε να αλλάξουν και οι τροχοί, να υπάρξουν ενιαίοι τροχοί αυτή είναι μια δραστηριότητα που έχει εφταπλάσιο κόστος από την ίδια την αντικατάσταση του βαγονιού. Και μετά βέβαια έχει να κάνει και το κόστος χρήσης των βαγονιών με τον όλο υπολογισμό. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητα στο συντηροδρομικό τομέα βεβαίω, όπω είπαμε, θα οδηγούσε στο να προτιμηθούν οι οδικέ μεταφορέ. Δηλαδή ένα τρένο με 40 βαγόνια ισοδυναμεί με 60 με 60 φορτηγά, ακόμη και αν χρειάζεται να διασχίσουν πόλεις. Εδώ Μιλάμε για μια δυναμική αγορά φυσικά ως προς τα μεγέθη της, ε, την ε, ε, οδική δηλαδή, την αυτοκινητοβιομηχανία. Στη συνδρομικό δίκτυο και τα πράγματα είναι αρκετά ίσχα και σταθερά προς στιγμή. Τι προκύπτει από όσα μόλις σας εξέθεσα. Ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα μετά την παρουσίασή μου. Βάσει της Λευκής Βίβλου της ε, Επιτροπής, της Λευκής Βίβλου για τις Μεταφορές, ένας από τους στόχους ήταν να έχουμε τουλάχιστον 30% οδικών μεταφορών. Αλλά αυτό έχει ψηλό κόστος και θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων. Διερωτώμε, λοιπόν αν είναι επιτέξιμος αυτός ο στόχος, αν είναι εφικτός. Οι συνδρομικές μεταφορές θα υποστούν, ε, θα πρέπει να αναλάβουν αυτό το υψηλό κόστος για να προσαρμοστούν και άλλη απορία. Ίσως να μην χρειάζεται να ακολουθήσουμε μία ομοιόμορφη προσέγγιση για όλους που όμως να αντίκειται στα επιμέρους συμφέροντα των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα ελαφρώς. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητή τώρα ο κύριος ε, ε, Τόμας Μακάλουμ, ε, καθηγητής στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Good afternoon. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Θα, πρέπει να... θα ήθελα να σας μιλήσω για το θόρυβο από την αεροπλοεία. Ξεκινάμε. Όπως ξέρετε, η αεροπλοεία έχει σημαντικό ρόλο στις... στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Τα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη αναπτύσσονται ανάλογα με τη ζήτηση. Και οι προβλέψει δείχνουν ότι η ανάπτυξη αυτή θα συνεχιστεί τι ερχόμενε δεκαετίε. Η αεροπλοεία επηρεάζει ήδη χιλιάδες στις ζωές τους. Χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε καθημερινή βάση. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι μοιάζει τα προβλήματα του θορύβου να χειροτερεύουν στο μέλλον. Αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία, στην, ε, στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και όσοι είναι πιο ευάλωτη στις διαταραχές από τους θορύβους των αεροσκαφών, περισσότερο από άλλες μορφές μεταφορών, αυτό έχει να κάνει περισσότερο επειδή τα αεροσκάφη μπορούν να περνάνε πάνω από το σπίτι σου ας πούμε και να φοβάσαι ακόμη και ότι έχεις να βρεθείς τυχαία στο δρόμο μιας πτήσης. Υπάρχουν ατυχήματα ατυχήματα γύρω από τα αεροδρόμια και αυτά αυξάνονται μάλιστα όσο πιο ευαίσθητος είναι ο κόσμος. Το μελετούμε το πρόβλημα από χρόνια κιόλα στο Μάντσεστερ και διαπιστώσαμε ότι ένα μεγάλο μέρος των ε, ευρωπαϊκών αεροδρομίων έχουν πολλούς περιορισμούς. Κλείνουν τα βράδια, έχουν περιορισμούς στη λειτουργία τους και όταν τα αεροδρόμια φτάσουν ε, το φουλ των δυνατοτήτων τους, Χρειάζεται βελτίωση στις υποδομές τους με νέα, νέους σταθμούς, νέα τερματικά, με νέες εγκαταστάσεις και βελτίωση. Τα μεγαλύτερα δρόμια στην Ευρώπη, μάλιστα, είναι αυτά που βρίσκονται ε, πιο κοντά στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πληθυσμού. Μοιάζει τα προβλήματα του θορύβου να μην πρόκειται να βελτιωθούν μάλιστα θα χειροτερέψουν γύρω από κάποια αεροδρόμια, κυρίως αυτά που αναπτύσσονται γοργά, διότι ο ρυθμός ανάπτυξης αυτής, αυτού του μηχανικού κλάδου είναι γοργότερος από τις τεχνολογικές εξελίξεις της ίδιας και το κατά πόσο προκύπτουν. Δηλαδή θα εκτίθενται ολοένα και περισσότεροι στο θόρυβο και θα υπάρχουν ολοένα και περισσότερα επεισόδια θορύβου. Καθώ χτίζει κανείς καινούργιες υποδομές, όπως ε, του διαδρόμου απογείωση ή του χώρου των αεροδρομίων, του αναδιερθρώνει για να αντιμετωπίσει τι απαιτήσει, τι δυνατότητε και τη ζήτηση, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη έκθεση των ευαίσθητων πολιτών στον θόρυβο. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονό ότι αλλάζει και η στάση των ανθρώπων. Δηλαδή, επίπεδα θορύβου που θεωρούνταν αποδεκτά στο παρελθόν, τώρα δεν θεωρούνται έτσι διότι ο κόσμος και περισσότερο ε, συμμετέχει ε, σε αυτές τις δραστηριότητες και έχει και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Το ίδιο και με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί και πιο ε, έντονα. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση να εκφραστεί όντως η αντίθεση προς την εξάπλωση των αεροδρομίων, προς την ανάπτυξή τους. Ακούσαμε και είδαμε και από άλλου ομιλητέ ότι συνέπειε από την έκθεση στο θόρυβο, δεν θα τι απαριθμίσω όλε, αλλά τα βασικά στοιχεία, και τα κρίσιμα στοιχεία φαίνεται να είναι επιπτώσει στην υγεία, διαταραχέ στον ύπνο, οι για την μάθηση στα σχολεία και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ε, υποφέρει από την γενικότερη όχληση, από τον διαρκή θόρυβο στο ε, γενικότερο περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί οι παράγοντε όχληση οδηγούν στι διαρκείς διαμαρτυρίες και τα παράπονα, καθώ και την αντίθεση στην ανάπτυξη και την επέκταση τη ε, αεροπλοεία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ε, βλάβες στην υγεία, με διαταραχές ύπνου, με διαταραχές μάθησης. Όλα αυτά σχετίζονται, όπως είδαμε με την έκθεση στο θόρυβο. Όμως η όχληση το γεγονό ότι η αντίληψη για το τι είναι αποδεκτό επίπεδο θορύβου επηρεάζεται, αυτό έχει να κάνει με παράγοντες που πολλές φορές δεν έχουν σχέση με τις ακουστικές ε, δυνατότητες, με την ακουστική πρόσληψη και αλλάζουν και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτά τα ζητήματα είναι που οδηγούν σε παράπονα και προσφυγές και διαμαρτυρίες. Τα ζητήματα αυτά, καθε αυτά, μετριάζονται από κάποιους παράγοντες μη ακουστικούς. Συγγνώμη. Α, να. Δηλαδή, εάν θεωρεί κανείς ότι ενοχλείται ή όχι, ε, αυτό εξαρτάται από τους μη ακουστικούς παράγοντες, όπως έλεγα. Τον τρόπο ζωή του δηλαδή. Αν ζει περισσότερο εντός του τι κατοικίε του ή όχι. Εάν ζει στην εξοχή σε ένα προάστιο ή σε ένα αστικό κέντρο. Εξαρτάται από το πόσο πλούσιο είναι κανεί, πόσα χρήματα έχει. Εξαρτάται αν είναι ιδιοκτήτη του σπιτιού που κατοικεί. Εξαρτάται από το εάν φοβάται τα αεροπορικά τυχήματα ή όχι. Εάν φοβάται επίση ότι θα επηρεαστεί η τιμή ε, του σπιτιού που κατοικεί από το αεροπλάνο που περνάει. Οι έρευνε που διεξάγαμε δείχνουν ότι οι άνθρωποι φοβούνται κυρίω για το μέλλον. Διότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι ζωές μας έχουν αλλάξει δραματικά και ο κόσμος κοιτάζει τι θα γίνει και σε άλλα δέκα χρόνια και φοβάται πώς θα είναι τότε η ποιότητα ζωής του. Επηρεάζεται επίσης από το αν κανείς έχει κάποιο όφελος άμεσα από το αεροδρόμιο. Αν δουλεύει κανείς ένα αεροδρόμιο, ε, το ανέχεται. Εάν όχι, γιατί να ανεχτεί τις ε, οχλήσεις που προκαλούνται. Οι έρευνες δείχνουν ότι 30% της όχλησης έχει να κάνει με τον ίδιο τον θόρυβο 30% έχει να κάνει με τους μη παράγοντες και άλλο ένα 30% είναι οι ατομικές ε, αντιλήψεις που έχει ο καθένας. Ξέρουμε ότι κάποιοι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι ή ευαίσθητοι, ενώ άλλοι όχι. Επίση, βλέπουμε εδώ δύο διαφορετικά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω σε αυτά τα κουτάκια. Ένα είναι η έκθεση στο θόρυβο και το άλλο είναι η απόκριση του κόσμου στι πηγέ θορύβου. Το πρώτο, όπω θα μπορούσε να πει κανεί, έχει να κάνει με τα ίδια αεροσκαφών, με τον αριθμό των πτήσεων, τι ε, χρονοθυρίδε τη ημέρα και το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη και του μη ακουστικού παράγοντε που επηρεάζουν την αντίληψη, όπω είπα. Η έκθεση στον θόρυβο ε, μετράται με συγκεκριμένα συστήματα παρακολούθηση και συγκεκριμένα μοντέλα, όπω ε, είπα προηγουμένω, ενώ οι στάσεις του κόσμου με μελέτες, με διαβουλεύσεις και με τι ε, παράπονα έχουμε συγκεντρώσει. Ο τρόπος για να ελεγχθούν όλα αυτά αλλάζει επίσης πάρα πολύ από μέρος σε μέρος. Δηλαδή υπάρχει ένα ρυθμιστικό σύστημα, μια ρυθμιστική προσέγγιση στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ έκθεσης στο θόρυβο και τις στάσεις που μπορεί κανείς να τηρεί ασχέτως με την έκθεση προβλέπει το γεγονός ότι υπάρχουν ε, διακυμάνσεις στην αντίληψη και τη στάση των ανθρώπων γύρω από τα διάφορα αεροδρόμια στην Ευρώπη, την ποιότητα της ζωής τους, το προσδόκιμο ζωής, το κατά πόσο έχουν συμμετοχή στα κοινά και το καθεξής και υπάρχει και ένας βαθμός ελαστικότητας, δηλαδή ο θόρυβος μπορεί να αντιμετωπιστεί σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων δράσης κατά του θορύβου τα οποία μπορεί να έχουν βασιστεί σε δημόσιες διαβουλεύσεις και να έχουν ληφθεί και ανάλογες προβλέψεις ε, για την καταλήξη κανείς αυτής της αποφάσης. Αλλά η ρυθμιστική προσέγγιση αναγνωρίζει πρέπει να υπάρξουν και όρια, όπως είπα προηγουμένως. Όρια στην προστασία της υγείας, ε, όρια στην προστασία του ύπνου ε, και σε κάποιες περιπτώσεις και στην προστασία της παιδείας. Ανάλογα με την αρχή της επικουρικότητας επίσης, αυτή η ρυθμιστική προσέγγιση ε, προωθεί και τη σωστή χρήση γης, το σχεδιασμό χρήσης γης για να προστατεύσει τον κόσμο από το θόρυβο. Αλλά αυτό θα ανέφερα και αργότερα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε λοιπόν είναι ότι τα αεροδρόμια είναι ακίνητα ε, περιουσιακά ε, στοιχεία. Ε, τα αεροσκάφη μπορούν να μετακινούνται, τα αεροδρόμια παραμένουν και δεν μετακινούνται. Είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμό των αεροδρομίων στην Ευρώπη που μετακινήθηκαν, όπω του Μονάχου τη Αθήνα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι, διότι δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα λίγο παραπέρα. στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμα καμία τέλεια λύση τακτική. Δεν μπορεί να γίνει ένα αεροσκάφο απολύτω αθόρυβο. Οπότε πρέπει να ε, υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση. Προσέγγιση που θα κάνει διάκριση μεταξύ τη έκθεση στο θόρυβο και τη στάση του κόσμου. Ε, την αντίληψη που έχουν. Πρέπει να προσαρμόσουμε τα όρια και του στόχου μα για την προστασία τη υγεία, τη του, για να προστατεύσουμε τον ύπνο και την παιδεία και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό, όπω εδώ προτείνω. Ε, παράλληλα όμω πρέπει να δούμε και πώ θα επηρεάσουμε τη στάση του κόσμου. Δηλαδή είναι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια τα ευρώ που δαπανώνται για να μειώσουμε την έκθεση στο θόρυβο ε, κατά έναν δεσιμπέλ ένα αεροσκάφος. Ε, αυτό δεν χρειάζεται τόση προσπάθεια. Η μόνη αξία αυτής της προσπάθειας έχει να κάνει με τους κανόνες του ΙΚΑΟ που ε, θα επιτρέψουν την πιστοποίηση των αεροσκαφών εν τέλει. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει καλύτερη τεχνολογική και επιχειρησιακή αξιοποίηση των όσων διαθέτουμε για να μπορεί και ο κόσμος να τα ε, καταλάβει, να τα προσέξει και να τα δεχτεί. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε τους ακουστικούς παράγοντες. Να ορίσουμε κατά πόσον ο κόσμος ε, οχλείται όντως ή το φαντάζεται. Επίσης πρέπει να υπάρξει δράση από τα ίδια ώστε να προωθήσουν την ανοχή στο θόρυβο, ε, εκεί όπου δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό χρειάζεται εκστρατείες ε, ενημέρωσης, χρειάζεται όρια για την εχορύπανση ή τέλο πάντων ε, να στείλει κανείς γράμματα στον κόσμο που να λένε ότι όσο αναπτυσσόμαστε και επεκτηνόμαστε θα σας προστατεύουμε παρόλα αυτά. Δηλαδή να δώσουν λόγο στις διάφορες κοινότητες αεροδρόμια να ανέχονται το θόρυβο και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και αποζημιώσεις για να μπορεί ο κόσμος να μετακομίσει. Όλα αυτά θα ωφελήσουν μόνο και μόνο τα ίδια τα αεροδρόμια διότι πρόκειται για επιχειρήσει που θέλουν να αναπτυχθούν. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει τα αεροδρόμια σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξη. Πώ μπορεί να αναλάβουν τέτοια δράση τα αεροδρόμια. Για να πάμε λοιπόν παραπέρα. Πρέπει να ξαναδούμε τα όρια για την έκθεση στο θόρυβο για την προστασία τη υγεία. Χρειαζόμαστε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να αντισταθμίσουμε τα κενά ανάπτυξη. Πρέπει να κάνουμε έρευνα για του μη ακουστικού παράγοντε που επηρεάζουν τη τάσει του κόσμου. Επίση, χρειάζεται πραγματική συμμετοχή του πληθυσμού και των πολιτών στην ανάπτυξη των αεροδρομίων και χρειάζεται τα αεροδρόμια να ε, γίνουν χώροι ευχάριστοι γύρω από αυτά να μπορεί να κατοικεί ο κόσμο και μάλιστα ευχάριστα. Ε, τότε θα μπορέσουν πραγματικά τα αεροδρόμια να αναπτυχθούν και να προσφέρουν τη συμβολή του στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Κουραστικές οι τέσσερι αυτέ ομιλίε Τώρα ακολουθούν οι ερωτήσεις. Η Γκέζινε Μάης είναι πρώτη αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις και τελευταία ε, ε, ε, κάλεσε μια ερώτηση. Είπε ο κύριος Καλούμ ότι υπάρχει και ένα υποκειμενικό στοιχείο από το θόρυβο. Δεν είναι τόσο αντικειμενικό. Αυτό δυσκολεύει και την πολιτική λοιπόν. Και ρωτώ και τους προηγουμένους που μιλήσατε για την επιβάρυνση από το θόρυβο. Αυτό πώς το μετράμε σε δεσιμπέλ ή σε αντίληψη του κόσμου ότι με ο θόρυβος. Γιατί ακούσαμε ότι πάνω από 70% ε, των ανθρώπων υποφέρουν από το θόρυβο στον αυτοκινητόδρομο, εντάξει και λιγότερο από το σιδηρόδρομο και την ε, αεροπορία. Ε, αλλά είδαμε και μια διαφάνεια που έλεγε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τους ενοχλεί ο θόρυβος. Πώς διατυπώνεται η ερώτηση. αυτό το πράγμα το μετράμε. Ε, είναι η αίσθηση της ενοχλής από το θόρυβο και ρωτάω και τον κύριο Τόμας. Ε, έχω ακούσει επανειλημμένως διάφορα πράγματα από αερομεταφορείς, από εταιρείε που, ότι δεν επιτρεπόταν να περνάνε πάνω από κατοικημένες ε, περιοχές γιατί ενοχλούσε τον κόσμο. Παρόλο που ήταν τέτοια η απόσταση από το έδαφος των αεροσκαφών όταν περνούσαν πάνω από την πόλη που αποκλείεται να του ενοχλούσε ο θόρυβο. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια, ένα ψυχολογικό στοιχείο εδώ στην πολιτική. Υπάρχει νευρο, νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Μπορείτε να πείτε ότι είναι καλός ο θόρυβος από τα αεροπλάνα γιατί φέρνουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και τότε θα χαρούνε, θα είναι μουσική, δεν θα είναι θόρυβος. Ε, βέβαια, είναι δύσκολα αυτά τα ψυχολογικά. Ε, προηγουμένως ακούσαμε ότι 40 δισεκατομμύρια είναι λέει το ετήσιο κόστος ε, που προκαλεί ο θόρυβος ε, στην Ευρώπη. Πόσο θα κόστιζε ε, να έχουμε μέτρα μείωσης του θορύβου. Κόστος ωφέλεια λέγεται αυτό. Και ένα τρίτο και τελευταίο ερώτημα. Έχετε υπολογίσει την ηλεκτρονική κινητικότητα στον αυτοκινητόδρομο. Την ηλεκτρική, συγγνώμη, αν είναι ηλεκτροκίνητα τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ, η κυρία Λουκασεύσκα. E, Άκουσα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τις παρεμβάσεις και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή Χέστον, ο οποίος τόνισε την χρήση των ε, διαφόρων μορφών και τεχνικών πέδησης. Πιστεύω ότι αν υπάρξει κάποια νομοθεσία στον τομέα αυτό θα πρέπει να βασιστούμε στην ανάλυση της πραγματικής κατάστασης. Δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε μόνο σε παρατηρήσεις όπως ε, ότι κάποια κράτη-μέλη έκαναν ε, εφαρμογή δίχως να λάβουμε υπόψη ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για, την, ε, τον χώρο. Και ε, πρέπει να κοιτάξουμε το πώς θα επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων κλάδων και ούτω καθεξής. Και στην ουσία μπορεί και να μην έχουμε περιορίσει την χορύπανση. Εξάλλου είναι αδύνατον να περιορίσουμε τον, ε, τον θόρυβο εντελώς η, ε, η χορύπανση από τους την οδική κυκλοφορία ή από τη συνδρομική εντάξει, είναι μία μέθοδος θα είναι να απομακρύνουμε τους αυτοκινητοδρόμους και τις ιδιοτροχές από κατοικημένες περιοχές. Φυσικά τονίσατε ότι ο μεγαλύτερη χορύπανση προκαλούν οι αυτοκινητόδρομοι, οι οδικές μεταφορές. Θα πρέπει ως εκ τούτου να μειώσουμε την ε, μεταφορές εμπορευμάτων και όχι μόνο οδικός και να μεταφερθούν στην ε, σιδηροδρόμους. Φυσικά δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω πως όποιες λύσεις προβλέπει η οδηγία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και ελπίζω να βασιστούν σε ακριβή στοιχεία και σε αξιόπιστα. Είμαι επίσης της γνώμης ότι θα ληφθούν υπόψη και οι γνώμες των προσκεκλημένων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Πρόσφατα διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο σε μια εφημερίδα ότι ο θόρυβος στον αυτοκινητόδρομο χειραγωγείται. Στην έγκριση των ε, τύπων είναι 74 ε, τα δεσιμπέλ στα αυτοκίνητα και 80 ε, στις μοτοσικλέτες. Αλλά αντίστοιχα με το Dieselgate αυτό είναι μόνο στο εργαστήριο, ας πούμε, τηρείται. Σε πραγματικές ε, συνθήκες ε, απέχουν πάρα πολύ και πέρα από τα πρότυπα τα αυτοκίνητα τελικά εκπέμουν τετραπλάσιο θόρυβο. 12 δεσιμπέλα έλεγε η Mercedes, διπλασιασμό, BMW 72 ήταν τετραπλάσιο από ότι στο τεστ και η Ducati ήταν τριπλάσιο. Τι, που, τι φταίει, υπάρχει ένα τρίκ, ένα σύστημα ε, στην εξάτμιση με κάτι βαλβίδες. Και σε κάποιες περιπτώσεις ε, η βαλβίδα εξουδετερώνεται και είναι πιο δυνατός ο θόρυβος. Τα λέει αυτά η αυτοκινητοβιομηχανία, είναι όλα νόμιμα γιατί δεν απαγορεύεται στο θόρυβο να γίνεται αυτό. Ερώτηση, αυτό το έχετε ακούσει εσείς. Έχει γίνει κανένα όρυβο σχετικά και τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μην έχουμε και ένα ε, ε, noise gate μετά το diesel gate. Μετά, ε, καταπολέμηση του θορύβου στην πηγή. βεβαίω είναι αυτό αποφασιστικό, αλλά και εκεί είναι θέμα τιμής. Ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, θα θέλαμε 12 δισεκατομμύρια για την ε, προστασία από το θόρυβο. Αυτούς τους τείχους που βάζουμε στις αυτοκινητοδρόμους. Αν πάμε όμως στο διασυναριακό εμπόριο, στις εμπορευματικές μεταφορές με το τρένο, χρειάζεται μόνο 1,5 δισεκατομμύρια. Ε, είναι πιο αθόρυβο, είναι πιο γρήγορο και θα εξοικονομούσαμε και 10 δισεκατομμύρια. Είδαμε πρόσφατα στην Τσεχία ε, τέτοιες ε, παριές ε, και εγώ δεν θέλω να μένω ή να είμαι σε ένα τρένο που να έχει γύρω-γύρω τύχη. Εγώ είμαι από το Βερολίνο και έχω ζήσει το τείχο που ήταν 3 μέτρα και 60 και τώρα χτίζουμε τείχη για την προστασία του θορύβου 6 μέτρων. Είναι τρέλε αυτά τα πράγματα, είναι παραφροσύνες. Είναι τρομερές ε, επενδύσει και όχι η καταπολέμηση του θορύβου στην πηγή. Και η βιομηχανία στέλνει στην Ευρώπη πιο αθόρυβα τρένα, σερμούς από ότι εδώ ή στη Γερμανία δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα, είναι πολιτική βούληση, γιατί είναι πιο αυστηρή νομοθεσία στην Ιαπωνία Εκεί το τηρούνε. Εδώ τίποτα. Αντίστοιχα με τις εκπομπές στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, στα πετρελαιοκίνητα ήταν πιο αυστηρές οι προδιαγραφές, γι' αυτό ήταν καλύτερα τα αυτοκίνητα και τους εξαπατούσαν και καλύτερα και πάει λέγοντας. Οι Ελβετοί το έχουν καταλάβει, έχουν ε, πει απαγορεύεται από το 2020 και μετά. Και τώρα βγαίνει η πολωνική ε, αερομηχανία που παράγει σειρμούς για εμπορευματικέ μεταφορές και ο διάδρομος ε, Ρότερνταμ-Γένοβα είναι ο πιο σημαντικός ε, και καταργηθούν αυτά γιατί θα τα απαγορεύσει η Ελβετία, τότε βλέπετε τι συμβαίνει. Τα είπε και ο κύριος Χέχτ και ποιος υπαγορεύει τις εξελίξεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τσακωθήκαμε καιρό και είπαμε 260 εκατομμύρια έχουμε για να αποσυρθούν τα παλιά βαγόνια και να βελτιωθούν και μέχρι 20% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Έγινε μεγάλος καυγάς, αυτό πέρασε, άρα ορισμένα κράτη και ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρείες δεν το αξιοποιούν αυτό, δεν το εκμεταλλεύονται. Αυτή δεν θα ήταν η σωστή λύση. Θυμίζω πώς αντιλαμβάνεται κανείς το θόρυβο στη Γερμανία προσέφυγε κάποιος γιατί λέει παίζουν παιδιά το μεσημέρι, το μεσημέρι έτσι, μία με τρεις ε, στην παιδική χαρά παιδιά και κάνουν φασαρία. Και ήθελε λέει να κλείνει η παιδική χαρά μία με τρεις και όταν έκανε την καταγγελία αυτή. Ευτυχώς δεν πέρασε. Αλλά αν είναι αυτό το πρόβλημα και αγνοούμε το αυτοκινητόδρομο, το αεροπλάνο και το σιδηρόδρομο, τι να πει κανεί, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και τελευταίο, ακούσαμε ότι στην Πολωνία είναι επταπλάσιο το κόστος εξυγίανσης ε, των σειρμών. Νομίζω δεν είναι ακριβώς αυτό, έχω άλλη πληροφόρηση εγώ. Αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό. Στην Πολωνία δεν έχουν διόδια ε, στον αυτοκινητόδρομο. Στη Γερμανία κάθε μηχανή για κάθε χιλιόμετρο τρένου ε, θα πρέπει να πληρώνει ένα τέλος, ένα διόδιο. Ε, αν είναι τεχνητά φτηνό ο αυτοκινητόδρομος και τεχνητά ακριβώς ο σιδηρόδρομος, δεν έχει καμία πιθανότητα να επιβιώσει το τρένο. Θα μπορούσαμε να το δούμε και από πλευρά τιμολόγηση και, και ένα οικονομικό κίνητρο να ε, εξυγχρονιστούν οι σειρμοί. Αν υπάρχει βούληση, αν υπάρχει θέλω, υπάρχει και μπορώ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα ανυπέρβλητα εμπόδια. Αυτά. Ζήτησε το λόγο συνέφηση από την Πολωνία. Ja tylko odpowiadając na Θα ήθελα να απαντήσω στον Πρόεδρο, ο οποίος διερωτάται πώς είναι το ψηλό το κόστος για την Πολωνία. Διότι στην Πολωνία έχουμε ε, διαφορετικούς τροχούς για την εγκατάσταση λοιπόν αυτών των, ε, των συστημάτων πέδησης ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο ακριβό να επιτευχθεί χρειάζεται ω εκ τούτου να τηρηθούν κάποια πρότυπα, κάποια στάνταρ. Σε ό,τι φορά όμω το παλιό ε, υλικό, το συνδρομικό, το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, εάν θελήσουμε να εγκαταστήσουμε νέους, νέους τροχούς στα βαγόνια, τότε θα κοστίσει πολύ, πολλά χρήματα. Εντάξει, να το απαντήσουν. Ε, θέλω να πω και κάτι που ακούσαμε σήμερα το πρωί. Στη Φιλανδία και στη Σουηδία ε, δεν επιτρέπεται να βάλουν αυτά τα σύνθετα υλικά, συστήματα πέδησης στα τρένα γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί ε, από τον πάγο δεν φρενάρουν τα τρένα. μπορεί να κάνει ναι, λιγότερο θόρυβο, είναι πιο επικίνδυνο. Ο κύριος Σέμπερλε, απάντηση πρώτη. Για την πρώτη ερώτηση. Ε, ο ήχος ε, μετριέται. Αυτό είναι φυσική. Ο θόρυβος είναι υποκειμενικό. Ρωτάς αν σε ενοχλεί ο θόρυβος. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Ήχους μετράμε. Και η αντίδραση στον αυτοκινητόδρομο τα τελευταία χρόνια και στο σιδηρόδρομο παραμένει αρκετά σταθερή. Σε μια ερώτηση πόσο σας ενοχλεί το τρένο. 60 ε, δεσιμπέλα ας πούμε, είναι το ποσοστό του πληθυσμού. Και το τι είναι υποφερτό και τι δεν είναι, θέμα ιδιοσυγρασίας. Τα άλλα πράγματα, η μέτρηση των θορύβων, μάλλον των ήχων, είναι φυσική. Ο θόρυβος είναι υποκειμενικό συνέστημα. Τώρα, αν έχεις δυσκολίες και ενόχληση στην επικοινωνία, στον ύπλο, ε, αύξηση του κινδύνου ε, εφράγματος, αυτό ε, είναι μετρήσιμη μεγέθη. Ε, τώρα, τα αποτελεσματικά μέτρα. Εγώ δεν έχω 40 ε, δισεκατομμύρια ε, για την καταπολέμηση του θορύβου στην πηγή, 10 δις στη Γερμανία. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι, για να το πω απλουστευμένα, όσο πιο νωρίς αναγνωρίζει κανείς το σχεδιασμό το πρόβλημα του θορύβου, τόσο πιο εύκολο είναι και πιο φτηνό πρόληψη. Ε, στον αυτοκινητόδρομο, δύο μέτρα σκέφτομαι, το βασικό πρόβλημα είναι όταν περνάνε μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι μέσα από ο, κατοικημένες περιοχές μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα. Έχουμε τη ταχύτητα με 30 χιλιόμετρα. Το, βράδυ έτσι κι αλλιώς δεν καταραίει καμία κυκλοφορία, ούτε το πρωί. Σχεδόν δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα ε, το μέτρο. Μειώνεται ο θόρυβος ε, κατά 3 δεσιμπέλ. Ε, και Επίσης αυτό έχει να κάνει και με τα οδοστρώματα. Ε, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικές προοδοί τεχνολογικές και επιστημονικές. Μειώνεται ο θόρυβος ε, κατά 2-3 δεσιμπέλ ε, στις πόλεις. Δεν είναι πολύ ακριβό. 10% ίσως αυξάνεται το κόστος στην ασφαλτόστρωση. τώρα, για το θέμα της κινητικότητας ή ακινησίας, γιατί ακούμε και το επιχείρημα ότι το ελαστικό είναι εκείνο που προκαλεί το θόρυβο στο δόστρωμα. Ε, για την, όχι την ακινησία, την ηλεκτρονική κινητικότητα. Δηλαδή δεν φταίει ο κινητήρας για το θόρυβο, φταίει το λάστιχο ε, που φρενάρει στην άσφαλτο ή που προκαλεί το θόρυβο αυτό όταν τρίβεται στην άσφαλτο. Όταν μειώνεται ο θόρυβος, ε, στην ηλεκτροκίνηση έχει σημασία η ταχύτητα. Μέχρι το 2014 υπήρχαν πολλά τεχνάσματα και μεγάλη εξαπάτηση, αλλά για το θόρυβο δεν ξέρω και ορισμένοι λέγουν ότι συνεχίζεται αυτό. Ε, παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 να το ελέγξει και να κλείσει τα παραθυράκια στην νομοθεσία, διότι... Ε, υποτίθεται ότι είναι αθόρυβα τα αυτοκίνητα, αλλά τελικά ξυπνάνε τον κόσμο. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Sorry, sorry. Er Για τα 50 δεσιμπέλ και πόσο ενοχλεί ο θόρυβος. Αυτή είναι μια τιμή, τα 50 δεσιμπέλ, που είναι αρκετά υψηλός ο ήχος και καμιά φορά και 30 δεσιμπέλ. Εξαρτάται. Αν προσανατολιστούμε σε αυτή την τιμή θα έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Αν κάνουμε συζήτηση επί της αρχής, ποιος θα κάνει τι, θα χάσουμε δεκαετίες ξανά και θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Και θα γίνει πολύ στόρυβος για το τίποτα. Τα 55 δεσιμπέλα, ας πούμε, είναι κάτι το ενοχλητικό. Αν θέλει κάποιος ε, να αμφινταλατεύεται και να ολιγορήσει, αρχίζει τη συζήτηση αυτή την κολοκυθιά για τις τιμές. Τώρα, τα θέματα ε, του κόστους έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες. Στις εναέρειες μεταφορές, όταν κάποιος σχεδιάζει ένα αεροσκάφος, έχει πέντε τιμές. Ε, πόσες θέσεις θέλουμε να έχουμε, σε τι απόσταση να πετάει, πόση κυροζήνη να καίει το χιλιόμετρο, τι κόστος ε, έχει και τι θόρυβο κάνει και θα πρέπει ε, ο θόρυβος να, να ενταχθεί μάλλον στο κόστος ε, για, το σιδηρόδρομο, στο πολωνικό παράδειγμα. Αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε το σιδηρόδρομο, ε, τα τελευταία 15 χρόνια χάθηκε το, η μισή αγορά και μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατρακύλα, αλλά μπορεί να υπάρξει και καινοτομία στο σιδηρόδρομο που θα του δώσουν περισσότερα μερίδια αγοράς. Ας πούμε, κάποια φρένα, κάποια συστήματα πέδησης που από 50.000 ευρώ και πάνω ε, μειώνουν και το κόστος αλλά λύνεται και το πρόβλημα του θορύβου. Αλλά στην ε, Πολωνία ε, είναι 20 με 40 χιλιόμετρα οι αποστάσεις που διανύουν το χρόνο και τα συγκεκριμένα λάστιχα, μάλλον συστήματα πέδησης δεν βοηθούν. Και υπάρχουν ε, και άλλα ε, φρένα που ενεργειακά ε, είναι κάτι το οποίο είναι εκτός συζήτησης και οι Τσέχοι έχουν τέτοια συστήματα. Είναι το, σταδιακά φρενάρι, όχι απότομα ο σειρμός. Πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε κάπως διαφορετικά. Σκεφτόμαστε μόνο το κόστος, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί θα καταστρέψουμε και θα σκοτώσουμε κάθε μέτρο κατά πολέμηση του θορύβου. Συνοψίζω. Όσο προχωράνε οι τεχνολογίες, ε, μπορεί να είναι ουδέτερο ε, ως προς το κόστος το θέμα της καταπολέμησης του θορύβου ή ακόμα και φθηνότερο. Τώρα, τι γίνεται με τη συμπεριφορά συγκεκριμένων συστημάτων πέδησης το χειμώνα. Υπάρχει ε, ε, μια τιμή τριβή που όταν χαμηλώνει η ταχύτητα μπορεί να αυξάνεται. Ιδιαίτερα όταν έχουμε πέτρελαιομηχανές, ε, βαριά τρένα που πρέπει να τραβάνε και σειρμούς πολύ βαριούς, μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά το τρένο. Αν πω στην εταιρεία σιδηροδρόμο ότι θέλω ε, ε, όλα τα τρένα, όλοι οι σειρμοί να έχουν τα ίδια συστήματα πέδησης, θα αναβαγίσουμε, θα εκτροχιαστούμε για να το πω με όρους τρένου. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές για τις ανάγκες του κάθε σειρμού, γιατί υπάρχει διαφορετική ανάγκη φρεναρίσματος κάθε φορά. Αυτά. Και η Φιλανδία και η Σουηδία, ναι, την ξέρω πολύ καλά την κατάσταση και στη Βόρεια Φιλανδία. Δεν είναι ηλεκτροκίνητα τα τρένα, είναι μηχανές δίζελ, ασθενείς, πολύ βαριά τρένα γιατί μεταφέρουν ξυλία και η δυνατότητα ε, επέδυσης φρεναρίσματος αυτών των σειρμών είναι πολύ μικρή. Ε, και ε, με τα σύνθετα υλικά είναι δύσκολο να φρενάρει το τρένο, είναι τεχνικά χαρακτηριστικά και λόγω των χαμηλών θεμεσιών. Ε, ε, οι Ρώσοι όμως εδώ και 60 χρόνια το έχουν λύσει το πρόβλημα και στη Φιλανδία ε, μπορούν να κυκλοφορήσουν τέτοια τρένα, αλλά είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές οι τεχνικές. Για τη Σουηδία δεν τα ξέρω πολύ καλά και απέχω. Για τη Φιλανδία έχω τη λύση πάντως. Ορίστε. Ε, σιγά σιγά τα βρίσκουμε, άμα έχετε και τη λύση. Ε, ο κύριος Κρόλ. Δεν θα ήθελα να δοθεί εντύπωση πως στην Πολωνία δεν γίνεται τίποτα για την αντιμετώπιση της χορύπανσης των αντίων. Τα νέα βαγόνια έχουν ήδη συστήματα πέδησης ε, με υλικό το οποίο περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο. Το, νέο, το πρόβλημα αφορά τη χρηματοδότηση μιας ε, τέτοιας ε, προσπάθειας. Ε, από ό,τι γνωρίζω, αλλά μπορείτε και να κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί μόνο σε περίπτωση αλλαγής του συστήματος πέδησης, αλλά όχι αντικατάστασης των τροχών. Σε περίπτωση που υπάρξει μια υποχρεωτική οδηγία TSI για τα βαγόνια που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, αυτό ε, το κόστος θα ανέρχεται σε 80 με 90 εκατομμύρια ετησίως προκειμένου να προσαρμοστεί το όλο υλικό, το όλο τροχαίο υλικό σε αυτά τα νέα πρότυπα. Και δεν είναι μυστικό, μπορώ να το πω, ότι το εισόδημα είναι 7,5 εκατομμύρια από τους ε, συνδρόμους στην Πολωνία. Ναι, φυσικά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την χορύπανση, αλλά τα κονδύλια τα οποία μπορούν να χορηγηθούν για την καταπολέμηση αυτής της χορύπανσης είναι περιορισμένα και αυτό περιορίζει ως εκ τούτου και την ανταγωνιστικότητα των τρένων. Και υπάρχει κίνδυνος φυσικά ότι ένα μεγάλο κομμάτι ε, εμπορικών μεταφορών θα μεταφερθεί στις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Τόμας. Ευχαριστώ. Να επιστρέψω στην όχληση. Πριν από πολλά χρόνια παρευρέθηκα σε μια συνεδρίαση κοντά στο αεροδρόμιο του Βουκαριστίου που ήταν ε, κατοικούμενη περιοχή πριν ε, μπει η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ε, θετικό αυτό που έζησα εγώ, είναι ένα σύμβολο σύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο και το σχολίασα θετικά. Πέντε χρόνια μετά έγινα πραγματική Ευρωπαίοι και άρχισαν να παραπονιούνται για το θόρυβο του αεροδρομίου. Καλό βέβαια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Υπάρχει συζητητισμό. Όταν λαμβάνουμε αποφάσει για το πώ ε, σχεδιάζουμε του αεροδιαδρόμου, ε, του διαδρόμου απογείωση ή την επέκταση του αεροδρομίου, πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ των οικονομικών ωφελών για την πόλη και την περιοχή ε, που θα εγκατασταθεί το αεροδρόμιο και τι ανησυχίε των τόπιων, των κατοίκων. Δεν μιλώ μόνο για την υγεία, μιλώ για την όχληση διότι κάποιοι φωνάζουν και χαίρονται οι γειτονέ του. Δεν ξέρω πώ μπορεί κανείς να εξορροπήσει πραγματικά εδώ τη διαδικασία λήψη αποφάσεων με αυτήν την αστάθμητη αντίληψη. Ευχαριστούμε, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις, οι ερωτήσεις και απαντήσεις. Ολοκληρώνεται για σήμερα αυτό το θέμα. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, γιατί πολλά μέσα μεταφοράς για να έχουν μέλλον θα πρέπει να καταπολεμήσουν το θόρυβο, να είναι αποδεκτό το επίθετο. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Βασικά αυτό που λείπει είναι πολιτική βούληση. Βεβαίως, όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση, ανέφερθηκα προηγουμένως στα διόδια. Γιατί δεν έχετε διόδια, ας πούμε, στην Πολωνία και στο αυτοκινητόδρομο και τόσο υψηλή χρέωση στο σιδηρόδρομο. Δισεκατομμύρια ε, για τα φορτηγά. Ε, στη Γερμανία, στην Πολωνία θα ήταν λιγότερα, αλλά αυτό που χρειάζεστε θα τα βρίσκατε αν βάζατε διόδια στους δρόμους. Μην κοιτάμε μόνο το θόρυβο, λίγο ευρύτερο πεδίο να έχουμε για να εξασφαλίσουμε και την κινητικότητα, να προστατεύουμε και το κλίμα και την υγεία των ανθρώπων επίσης. Ολοκληρώνεται λοιπόν για σήμερα το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σας παρακαλώ καθίστε ή φύγετε, γιατί έχουμε και άλλο θέμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι τελείως διαφορετικό. Σήμερα είναι ανάμεσά μας κάποιος που ζει την τελευταία του συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ο κύριος Λεβέντε Μπόζακ που τέσσερα χρόνια ε, δούλευε καταπληκτικά και μας φεύγει τώρα. Απίστευτο, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να τον ευχαριστήσω θερμά για την καταπληκτική συνεργασία, πάντα με μεγάλη ικανότητα και επαγγελματισμό. Περάσαμε πολύ καλά, είχαμε και πολλή δουλειά. Δυστυχώς εδώ τελειώνει αυτό, αλλά για το μέλλον ό,τι επιθυμείτε, καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Καλή συνέχεια. Και έκλεισε το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Τώρα είναι εντάξει το μικρόφωνο. Είχε κλείσει προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ε, λάθος, το πάτησα κατά λάθος. Έχουμε τον κύριο Λουκ Βίλιμς και τον κύριο Γιάνν Μόλεμα καλέσει. Ο Λουκ Βίλιμς είναι απληρωτή Γενικό Γραμματέα του Μπενελούξ και ο Γιάνν Μόλεμα ε, επικεφαλής ε, του τμήματος εσωτερικής αγοράς Μπενελούξ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά έκαστος, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Πρόεδρε. Αποτελεί τιμή για μα που βρισκόμαστε εδώ ανάμεσά σα, στην Επιτροπή Μεταφορών. Βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από την έκθεση σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές και θα σας πούμε τα ευρήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της ε, έρευνάς μας. Θα σας μιλήσω για το περιεχόμενο. Μια σύντομη εισαγωγή στην ε, έννοια της Benelux, η σημασία της ε, των μεταφορών στο Benelux, μερικές ε, αποτελέσματα από την έκθεση και την, κάποιες ματιές στο μέλλον και μετά τα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα του Μπενελούξ ε, συνεχίζει να εφίσταται και είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια διακυβερνητική ε, ε, συνεργασία ανάμεσα στην Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Η οικονομική συνεργασία είναι η ουσία της Μπενελούξ και η περιφερειακή συνεργασία η οποία έχει καταδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια μπορέσαμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά και αποδοτικά. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά ε, συμφωνίες όπως το Σέγγεν και άλλες που έχουν υπογραφεί στο Λουξεμβούργο. Το 2012 τα, ε, οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να, να ε, υπογράψουν μια νέα συμφωνία Μπενελούξου και υπήρξε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών. στόχο είναι η εμβάθυνση της συνεργασία ανάμεσα στα τρία κράτη, αλλά και η ενίσχυση του πρωτοπόρου ρόλου που παίξαμε και συνεχίζουμε να παίζουμε στην Ευρώπη. Με τη νέα συνθήκη η συμφωνία δεν αφορά μόνο ε, οικονομικούς κλάδους, αλλά επεκτείνει στον τομέα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και την βιώσιμη ανάπτυξη και θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πέντε θεσμοί. Το σημαντικό είναι η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στον τομέα των μεταφορών και θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω ε, την εσωτερική αγορά. Κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω το άρθρο 350 της συνθήκης Μπενελούξου ότι οι χώρες Μπενελούξου θέλουν να προχωρήσουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της ιστορικής αγοράς τους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όμως να παρεμποδίσουν την δραστηριότητα των άλλων κρατών. Αυτό παρουσιάζει πλεονεκτήματα και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Τώρα. Να σου πω ότι υπάρχει ένα ελεύθερο καμποτάζ ανάμεσα αυτά κράτη. Τα φορτηγά μπορούν να κυκλοφορούν με φορτίο 44 τόνων αντί για 40 που στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2014 ο πρώην Υπουργός ε, κύριος Τίμερμανς υπέγραψε την απόφαση να ε, μπορούν αυτά τα φορτηγά να διασχίζουν τα σύνορα και επίσης υπογράφει συμφωνία για την ε, κυκλοφορία αυτών των ε, φορτηγών με μεγαλύτερο φορτίο ανάμεσα στο Βέλγιο και το... Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον συνάδελφο Μόλεμαν, ο οποίος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης που έχει γίνει. Μάλιστα. Λειτουργεί το μικρόφωνο βεβαίως. Ευχαριστώ Λουκ. Τα πρώτα ευρήματα ποια είναι αυτής της έκθεσης. Όπως λέει και ο τίτλος, οι μεταφορές δεν είναι ε, ουσιαστική σημασία μόνο για τον Πενελούξ αλλά και για όλη την εσωτερική αγορά όταν λειτουργούν σωστά. Θα τα δούμε αυτά στο επόμενο slide, στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε το θερμικό χάρτη της Ευρώπης. Ε, μας δίνει μερικές προφορίες. Πρώτα απ' όλα βλέπετε αυτές τις περιοχές στο κόκκινο ε, πάνω από τις χώρες Μπενελούξ που σημαίνει πολύ καυτή κυκλοφορία και βαριά εφοδιαστική δραστηριότητα σε μια σχετικά μικρή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δείχνει και η διαφάνεια ε, ποιες είναι οι πιο προσφυλείς ε, περιοχές ε, που θέλουν να εγκατασταθούν οι ξένοι επενδυτέ όταν έρχονται για να στείλουν τα εμπορεύματά τους όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η γενική εικόνα λοιπόν. Γιατί κάναμε μια μελέτη γι' αυτό ακριβώς το θέμα για τις εμπορευματικές ροές. Για διάφορους λόγους. Πρώτον, Ε, τα κράτη-μέλη μα, το Βέλγιο, οι κάτω χώρε και το Λουξεμβούργο και οι διάφορε περιφέρειες του Βελγίου ζητούν δράση. Βλέπουν ευκαιρίε και βλέπουν τι αγορέ να καινοτομούν περισσότερο και πιο γρήγορα από κάποιου κανονισμού, τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Ε, αυξάνονται οι εμπορευματικέ ροέ και αλλάζουν γρήγορα. Έχουμε νέα μέσα μεταφορών που εισάγονται και βεβαίω ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί όλα αυτά για να μα καθοδηγήσουν από ευρωπαϊκή πλευρά. Και επίσης όταν κάνουμε κανόνες, όπως ακούσαμε προηγουμένως, για τον Πενελούξ και την εσωτερική αγορά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα χρειαζόμαστε ε, κάποια στοιχεία και πληροφορίες για το πώς κυκλοφορούν τα εμπορεύματα στις χώρες Μπενελούξ και στις όμορες. Αν δούμε λοιπόν τώρα τα πρώτα μας ευρήματα, τι διαπιστώνουμε. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, για να δούμε, θα έρθει η διαφάνεια. Ωραία. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, της επικράτειας είναι μικρό. 1,7% είναι το Benelux ολόκληρη τη Ευρώπης από γεωγραφικού όρου. Είναι μικρή η επιφάνεια. Αν δείτε όμω ε, τι ροές των εμπορευμάτων ε, και το ΑΕΠ ε, που δημιουργείται είναι τριπλάσιο σε σχέση με την επικρατεία μας, 7,9%. Επίση, τι σημαίνουν οι συγκεκριμένοι τρόποι μεταφοράς ή τα μέσα μεταφοράς για το περιβάλλον των μεταφορών. Δεξιά θα δείτε και θα καταλάβετε την εσωτερική ναυσιπλοεία 78% ε, της ε, ευρωπαϊκής εσωτερικής ναυσιπλοείας εισέρχεται, εξέρχεται ή διέρχεται από τις χώρες Μπενελούξ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εμείς μπορεί να έχουμε κανόνες για τις χώρες μας για να προσπαθήσουμε να καινοτομήσουμε και να έχουμε μια ψηφιοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το Benelux πάνω από τρία τέταρτα της ε, Ευρώπης των προβλημάτων της. Ε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ να το μοιραστούμε μαζί σας αυτό το στοιχείο. Κάποια άλλα στοιχεία ακόμα. 24% επίσης ε, του ε, φορτίου του αερομεταφερόμενου φτάνει στην Ευρώπη μέσω των χωρών Βενελούξ και αυτό πολύ σημαντικό. Ε, θαλάσσιες μεταφορές πάνω από 20% του συνόλου, δηλαδή με διάφορα μέσα μεταφοράς, με αεροπλάνα και βαπόρια έρχονται εδώ πέρα τα εμπορεύματα, ήδη έρχονται και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, ε, τι άλλο βρήκε η έρευνα για να το εντάξουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τώρα ξέρουμε πάνω κάτω που είναι οι βασικές ροές ε, και ποια σύνορα περνούν. Ε, Κάτι που μας εξέπληξε και μας από τα ευρήματα είναι το εξή. Αν κοιτάξετε τις οδικές μεταφορές που είμαστε αρκετά δραστήριοι, αλλά σε αποφάσεις ad hoc κάθε φορά, τι βρήκαμε στην έκθεση, ότι 76 των οδικών μεταφορών ξεκινάει κάπου ε, που ξεκινάει από το Μπενελούξ μπορεί να περάσει κάποιο σύνορο, αλλά παραμένει σε μία από τις τρεις χώρες Μπενελούξ. Το 76%. Άρα θα μπορούσαμε να ε, νομοθετήσουμε ε, εντό Μπενελούξ για να ξεφορτωθούμε κάποιους φραγμούς και κάποια σύνορα και προβλήματα στα σύνορα. Αυτό ήταν το slide, η διαφάνεια που αναφέρεται σε αυτό που σας είπα μόλις. Αποτελέσματα και συμπερασμάτα. Τρίτα. Είμαστε ε, πρωταθλητές στην εφοδιαστική. Ε, το Λουξεμβούργο βγήκε δεύτερο, ε, τρίτη σε κατοχώρες και έκτο το Βέλγιο. Πάντως στο top 10 είμαστε στις 10 πρώτες χώρες. Βέβαια πρώτη είναι η Γερμανία, ο γείτονά μας, από το 2014. Αυτό δεν μας εκπλήσει. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη η περιοχή με μεγάλη δραστηριότητα οικονομική. Θα πρέπει και εφοδιαστική να είναι κρατεά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Τώρα πώς ε, μπορούμε να ανταποκριθούν αν αυξηθούν οι ροές, γιατί έτσι προβλέπεται, τουλάχιστον θα διπλασιαστούν, να μην πω ότι θα τριπλασιαστούν κιόλα μέχρι το 2030, άρα πρέπει να αναλάβουμε δράσεις έτσι ώστε να παραμείνουμε στις θέσεις αυτές τις ηγετικέ. Πώς αξιοποιούμε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνας. Βεβαίως, με ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, όχι μόνο στον Πενελούξ, αλλά και με τους εταίρους μας. Ε, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε σύνοδο και θα καλέσουμε και τους γείτονές μας. Κάνουμε πιλωτικά προγράμματα. Διάφορα τρέχουν ήδη, έχουν δρομολογηθεί για τις οδικές μεταφορές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, όπως είπαμε προηγουμένως, με βάση τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκής Ένωση, να υπάρξουν νομικέ συμφωνίε για να δημιουργηθεί ήδη μια εσωτερική αγορά Benelux και αργότερα ευρωπαϊκή για να διευκολυθούν ε, οι λύσει. και αν έχουμε καλές συζητήσει και αποτελέσματα από τα Υπουργεία μας μπορούμε γιατί όχι να το εξάγουμε αυτό και σε όλη την Ευρώπη προκλήσεις και προβλήματα που έχουμε παντού στην Ευρώπη, όχι μόνο στον Πενελούξ. Και αυτά τα μελέτησε η έρευνα. Και η έκθεση αυτή είναι προφανή. Έχουμε μαζικές ροές εμπορευμάτων στην επικράτειά μας και συμφόρηση. Εσείς το βλέπετε καθημερινά οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι στους δρόμους. Το ζείτε. Γύρω από τα μεγάλα λιμάνια και γύρω από τις μεγάλες πόλεις έχουμε μποτιλιαρίσματα και συμφόρηση. Θα πρέπει να έχουμε συνδυασμένες μεταφορές, να φύγουμε από ε, ένα μέσο μεταφοράς και να πάμε στο άλλο. Ποιο θα είναι αυτό θα δείξει. Οι στόχοι βιωσιμότητας απέχουν πόρο από τους επιθυμητούς. Ε, θα πρέπει να το δούμε και με την Ευρώπη. Η ψηφιοποίηση επίσης και ε, οι πληροφορικοί συστήματα FEE. E για την κυκλοφορία μπορεί να είναι τμήμα της λύσης. με ευφύ συστήματα, δεν λέω να αυξήσουμε τους δρόμους ή τις εσωτερικές έσοδους, αλλά και νέα μέσα μεταφοράς. Έχουμε νέους τρόπους πριν από 10 χρόνια. Κανείς δεν σκεφτόταν ότι θα μπορούσαν τα drones να χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές για παραδόσεις ε, εμπορευμάτων. Τώρα το ηλεκτρονικό εμπόριο οργιάζει ε, στις χώρες Benelux και ήδη κάποιες εταιρείες ε, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν drones για να παραδίδουν τα εμπορεύματα. Να πούμε και κάτι καλό για το τέλος. Μειώνεται και σταθεροποιείται η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Καλό είναι αυτό. Αλλά είναι εύθραυστη αυτή η εξέλιξη γιατί αναμένεται μεγάλη αύξηση των εμπορευματικών ροών. Αν δούμε τι θα γίνει στο προσεχές μέλλον, για τα δύο μεγάλα λιμάνια που είναι το Ρότερνταμ και η Αμβέρσα, το επόμενο διάστημα μέχρι το 2030 θα έχουμε 35, από 235 εκατομμύρια τόνους θα έχουμε 400 εκατομμύρια συγγνώμη, τόνους το 2030, από το 13 στο 30 και μάλιστα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει ε, ο τρόπος μεταφοράς από το Ρότερνταμ, να φύγουμε από τις οδικές μεταφορές, από το 55% να έχει πέσει το 35% για την Αμβέρσα, από 56% να, πέσει το 43% και να αυξηθούν οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές από το 35% στο 42%. Προφανές αυτό. Αυτό ισχύει επίσης και για το σιδηρόδρομο που θα διπλασιαστεί η χρήση. Κάποια πρώτα συμπεράσματα. Ίσως για να θυμάστε κι εσείς. Εμείς είμαστε ένα ζωντανό εργαστήριο για την Ευρώπη για να μελετηθούν καινοτόμε ιδέες, ιδέες που θέλουμε λίγο νωρίτερα να δοκιμάσουμε σε μικρή κλίμακα πριν επεκταθούν στην Ευρώπη, να το κάνουμε. Ε, για να ε, μάθουμε να διδαχθούμε από την εμπειρία τι λειτουργεί σωστά και τι λιγότερο. Και μπορούμε να είμαστε μια ταχεία οδός για τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια καινή πλατφόρμα για εφαρμογή ε, πολλών μέτρων και με πολλούς τρόπους. Είμαστε τρεις μάλλον μικρές χώρες, χώρες Benelux, Και με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύουμε συνήθως την νομοθεσία. Και ένα τελικό συμπέρασμα. Η επιτυχημένη συνεργασία Benelux στις μεταφορές ε, κρατάει την Ευρώπη σε κίνηση. Ε, σας ευχαριστώ ε, για τις, ε, την ευκαιρία που είχαμε να σας πάρουμε τις απόψεις μας και την ε, συζήτηση που ελπίζω να είναι γόνιμη. Ε, ανοίγει η συζήτηση. Ο Ζορς Μπαχ, καλό στα παιδιά. Όχι, ο Βιμ Βαντεγκάμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κοίταζα το Ζορς Μπαχ, γιατί είναι... Ε, έχει την πνευματική διοκτησία, κατέχει αυτού του, της να έρθει να παρουσιαστεί εδώ αυτή η μελέτη. Θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα διαβάσει αυτό το κείμενο και με εντυπωσίασε είναι αυτή που ονομάζουμε εμείς ε, γενική προσέγγιση, συλλογική, από ένα τμήμα της Ευρώπης που έχει συνολική εποπτεία ε, για την Ευρώπη. Του, του χρόνου θα πάμε στο Rail Baltica. Ε, όταν είσαι ε, Μπενελούξ και δρεύεις στις Βρυξέλλα, δεν έρχεται κανένας επίσκεψη, δεν έχει ταξίδι ε, μελέτης και αποστολή, μπορεί να έρθει όποτε θέλει. Πραγματικά πολύ ωραία αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το μέρος της Ευρώπης. Και έχω μερικές ερωτήσεις. Στην έκθεση, πώς να το πω τώρα, υπάρχει μια μικρή σύγκρουση με τη Βόρεια Ρινανία, Ρινανία-Βεστφαλία. Ε, είναι ένα ε, ένα τέταρτο άτυπο μέλος Μπενελούξ. Τι θα κάνετε, θα την συνδέσετε, όχι επίσημα λέω, έτσι τυπικά, ε, άτυπα, ουσιαστικά, ε, στις μεταφορές, στην πολιτική μεταφορών θα εντάξετε τη Βορεια Ρινανία Βεσφαλία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ε, το σύστημα διοδίων. Πάντα με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Η βελγική κυβέρνηση έχει ε, εισαγάγει ένα σύστημα διοδίων και ήταν πιο έξυπνη από την ε, γερμανική κυβέρνηση εδώ. Πιο έξυπνη με την έννοια την ε, Ολλανδική, όχι τη Γερμανική. Λογική δηλαδή λύση. Θα υπάρξει και ένα σύστημα διοδίων Βενελούξ γιατί υπάρχει βελγική προσέγγιση που οδηγεί σε προβλήματα στην Νότια Ολλανδία πλέον. Τώρα, η επίδοση και η παράδοση των δεμάτων. Έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Ρικέ, όπου έχουμε κάποια ελαφρά, ελαφρά οχήματα που παραδίδουν ε, δέματα και οι οποίοι δεν υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προσπαθούν να την παρακάμψουν. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι κάνουν αυτά τα ελαφρά ε, οχήματα που παραδίδουν δέματα. Έχετε κάποιες συστάσεις σε αυτό. Έχετε καμιά ανησυχία, σας προβληματίζει. Άλλο θέμα, Πρόεδρε. Το προσφυλές σας θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων Έχουμε περιφερειακά αεροδρόμια. Είναι θέμα του Κράμερ, αλλά το, το δανείζομαι. Ε, καλύπτουν το κόστο τους. Είναι βιώσιμα αυτά τα περιφερειακά μικρά αεροδρόμια. Αυτά προς το παρόν. Έχω κι άλλα, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, Ντομινίκ Νικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ενδιαφέρουσα ανακοίνωση θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση που εξαρτάται από την ερώτηση που έθεσε ο Βίδιαν σχετικά με τις ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις που έχετε με την Ρινανία Βεσφαλία καταλαβαίνω πως ε, ένα είδος ε, ενότητας ε, όγκου θα έλεγα θα ήθελα να μάθω εάν έχετε επαφές ή και σχέσεις με την περιοχή της Ότ που βρίσκεται ακριβώς ε, κάτω από την ε, στο υπογάστριο θα λέγαμε του Μπενελούξου και το κανάλι Σέντεξχο θα αποτελέσει για τις λιμένες του Βορρά σημαντική ευκαιρία θέτω το ερώτημα διότι ξέρουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί αυτή την κεντρική ζώνη της Ευρώπης ειδικά σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταφορές. Δεν πρόκειται για μια τακτική χρήση, αλλά η χρήση τους στην διεθνή μεταφορά. Ίσως θα έχω αργότερα κάποια ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα, Ζωσμπάχ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ε, συγχαρώ τους ομιλητές ε, στο πλευρό του κυρίου Κάμπ. Ευχαριστώ τους δύο κυρίους, πάρα πολύ καλή δουλειά τους, πάρα πολύ σημαντική. Τώρα απλώς ε, ακροθυγώς είδαμε τα θέματα, αλλά αν τα μελετήσουμε μπορούμε να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Για μένα είναι πολλά τα ερωτήματα που αναδύονται, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Βίμ Κάμπ το θέμα των διοδίων. Και επίσης, αν έχετε καμιά ιδέα για το πώς μπορεί να αναλυφθεί μια κοινή πρωτοβουλία. Και μια άλλη ερώτηση. Έχετε πάρα πολλά αριθμιστικά στοιχεία ε, για τους απασχολούμενους στον τομέα αυτό. Και από εκεί και πέρα, πώς μπορείτε να φανταστείτε μια συνεργασία ε, σε σχέση με τις αρμοδιότητες, μάλλον τα, ικανό, ε, τα προσόντα και τις ικανότητες και τις δεξιότητες. Υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ε, των πτυχίων των εργαζομένων. Ας πούμε στην εφοδιαστική έχω την αίσθηση ότι ο καθένας κάνει τα δικά του. θα μπορούσατε να σκεφτείτε καμιά ενιαία γραμμή για κοινή συνεργασία και τι γίνεται με τις υποδομές. Τώρα ε, υπάρχουν ε, πολλές προσπάθειες ανανέωσης των υποδομών για να ε, είναι η στόλη πιο φυσική προς το, φιλική προς το περιβάλλον, με τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου για την αυσιπλοεία και πάει λέγοντας. το έχετε σκεφτεί αυτό για τους κόμβους και την τη νέα μορφή μεταφορών. Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Τι γίνεται με τα γίγαν ε, liners, που αυτά τα τεράστια φορτηγά, τα μεγαθύρια των ασφάλτων. Τι γίνεται. 35% των συνδυασμένων μεταφορών ε, μεταφέρονται στο, στις οδικές μεταφορές γιατί είναι πιο φτηνό ε, από το σιδηρόδρομο. Δεν το θέλει κανείς, αλλά θεωρητικά ακούμε πάντα ότι άμα είναι μεγάλα κυκλοφορούν δύο φορτηγά αντί για τρία. Στη Γερμανία λείπουν 20.000 ε, θέσεις να παρκάρουν ε, στους αυτοκινητοδρόμους τα φορτηγά και αν μας έρθουν τέτοια μεγαθύρια πού θα τα βάλουμε. Ε, και βεβαίως κυκλοφορούν και πολλά άδεια γιατί, και ένα φορτίο γιατί είναι πάμφτινο. Στην Ελβετία δεν υπάρχει φορτηγό που να κυκλοφορεί άδειο γιατί είναι πανάκριβα τα διόδια και στις χώρες Benelux ε, υπάρχει διαφορά σε σχέση με ε, τις γειτονικές χώρες, καλά στη Γαλλία έχουν τελείως διαφορετικά διόδια. Ναι. Γιατί είναι τόσο μεγάλη η κυκλοφορία, επειδή δεν έχετε διόδια και δεν είναι μόνο τα διόδια φτηνά, είναι φτηνά και τα καύσιμα. Εγώ ξέρω πολλές εταιρείες φορτηγών που φεύγουν από την Ισπανία ε, φουλαρισμένοι, μετά πάνε στο Λουξεμβούργο και φουλάρουν γιατί είναι τόσο φτηνά, περνάνε τη Γερμανία και πάνε στην Πολωνία για να ξαναγεμίσουν. Δηλαδή κάνουν βόλτες στην Ευρώπη και πάνε και παίρνουν καύσιμο από εκεί που είναι πιο φτηνά. Αυτό ε, παραμένει ε, πλεονέκτημα, να είναι τεχνητά χαμηλή η τιμή της βενζίνης και να έχετε πολλή κίνηση. Και τι γίνεται με τους γείτονες. Εντάξει, γείτονες Γαλλία, Γερμανία στις χώρες Μπενέλοξ. Και η ε, δεν τολμάει να το αναφέρει πια. Βρυξέλλες Βαλανσιέν, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, μπορεί να μειωθεί κατά μία ώρα εάν για 800 μέτρα ξεχορταριάσουν τις ράγες για να πηγαίνει ο κόσμος με το τρένο. 800 μέτρα και θα μειωθεί κατά μία ώρα η διαδρομή τόσο τεράστιο πρόβλημα είναι και κάνουμε τεράστια παράκαμψη, πανάκριβη και σε χρόνο και σε χρήμα. Ε, δεν τολμάει πια να τα αναφέρει ο αυτά, αλλά από εκεί θα φύγουμε από το δρόμο και θα πάμε στο σιδηρόδρομο. Και τελευταίο παράδειγμα. Μια φορά το μήνα πολλοί εργαζόμενοι φεύγουν από τις Βρυξέλλες και πάνε Στρασβούργο. Αυτό το τρένο είναι καταστροφή σκέτη. Εγώ δεν το έχω πάρει ποτέ. Έχω ακούσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πέντε ώρες στο δρόμο, δεν έχει εστιατόριο, δεν έχει καφετέρια, καθυστερεί συνέχεια, δεν μπορείτε επιτέλους οι χώρες Μπενελούξ να το δείτε από κοινού και να πείτε ε, ότι θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και με τους γείτονες να το συζητήσουμε γιατί και ο Βιμ Βάντεν Βαντενκάμπ άκουμε λίγο, επειδή αναφέρθηκε στο Rail Baltica δεν σε αφήνω να μιλάς με το γείτονα, εγώ δάσκαλος είμαι γιατί μίλησε για το Rail Baltica θα πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα είναι κοινοπραξία τριών κρατών που είναι κυρίαρχα κράτη εδώ και λίγο καιρό αλλά συνδυάστηκε ε, για να φτιάξουν το Rail Baltica θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, υπόδειγμα κοινοπραξίας για το τρένο από Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, μπα και βρούμε την υγειά μας. Αυτά τώρα μπορείτε να απαντήσετε, παρακαλώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε και κύριοι για τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα ερώτηση για τη συνεργασία για τις περιοχές της περιφέρειας γύρω από την Μπενελούξ. Υπάρχει συνθήκη Μπενελούξ από το 2012 και μια πολιτική δήλωση μεταξύ των τριών κυβερνήσεων και την ε, κυβέρνηση της Βεσφαλίας στο Λουξεμβουργό την επόμενη φορά η Επιτροπή των ε, Υπουργών των Μεταφορών των Τριών Χωρών με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ρινανίας Βοσφαλίας θα συζητήσουμε ακριβώς αυτές τις συστάσεις με τη Ρινανία Βεσφαλία. Κύριε Ρικέ, για τη συνεργασία με τη Γαλλία στο επίπεδο των μεταφορών και στο επίπεδο των ε, οδικών διασυνδέσεων. Έχουμε αποτελεσματικότητα τη συνεργασία κατά του κοινωνικού dumping. Εξαιρετική συνεργασία δεν είναι παρόμοια με αυτή που έχουμε με τη Ρινανία Βεσφαλία βέβαια. Και σε ό,τι αφορά την, τα καύσιμα και την ε, τιμολόγησή τους, είναι από τα πιο σημαντικά θέματα, ζητήματα που απασχολούν τις χώρες Μπενελούξ. Γιατί είμαστε κλασική μορφή διασυνεργειακή συνεργασία, διακρατική και υπάρχουν και διαφορετικέ απόψει μεταξύ των τριών κυβερνήσεων. Ίσως να μπορούσαμε κάτι να δημιουργήσουμε από εδώ Μπενελούξ, αλλά υπάρχουν αποκλήσει απόψεων Ω ε, δημόσιοι υπάλληλοι που εργαζόμαστε για την Benelux, καταλαβαίνουμε ότι οι διαφωνίε ε, είναι κάτι το αναπόφευκτο, πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να βρεθεί και λύση. Θα τα συζητήσουμε και αυτά την επόμενη εβδομάδα. Για το σύστημα τιμολόγηση των οδικών μεταφορών. Για τα δύο όδια δηλαδή και το πώς αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε στην, Ολα... με την Ολλανδία, μεταξύ Λουξεμβούργου, Ολλανδίας και Βελγίου. Βεβαίω είναι σημαντικό να έχουμε βιώσιμες μεταφορές Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία σε κυβερνητικό επίπεδο. Και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι παρόμοια με όσα συζητιούνται και στο ε, Κοινοβούλιο. Και για την άλλη σας ερώτηση, και μετά θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο, στο Γιάνν Μόλεμα, για τα τεράστια φορτηγά, για τα κονβόι και το συνδυασμό φορτηγών με πολλά βαγόνια πίσω. Ναι, το 2014 ήδη είχαμε μια σχετική πρόταση στο Κοινοβούλιο. Έχουμε δύο αποφάσεις τώρα, δύο δηλώσεις μάλλον από τον Benelux για τα οχήματα των 45 στοιχείων. Ε, των 45 ποδών. Ε, εκεί βλέπουμε ε, κατά πόσον μπορούμε να εντάξουμε τα τεράστια φορτηγά αυτά, τα γιγαντιαία, τα τερατώδη φορτηγά όπως έχουν ονομαστεί. Και θα δούμε αν μπορούμε στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο να έχουμε κοινά προγράμματα. Δηλαδή από το αεροδρόμιο της Λιέγης υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρξει διασύνδεση με την Airlux και κάποιες εταιρείες επίσης ενδιαφέρονται να το χρησιμοποιούν τη νύχτα. Θα τα συζητήσουμε όπως είπα την επόμενη εβδομάδα σε επίπεδο υπουργών μεταφορών για να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις, αλλά σίγουρα υπάρχει μια διάθεση σε επίπεδο Benelux, μια όθηση για να χρησιμοποιήσουμε τέτοια δύο επιχειρήματα και να επιτελέσουμε πρόοδο. Στις κάτω χώρες, με τα μεγάλα, τα βαρέα φορτηγά είδαμε θετικά αποτελέσματα, ε, ήταν και χαμηλότερη συχνότητα όμως. Γιάννη, ναι, εάν δω τον κατάλογο, τα μικρά δέματα και η παράδοσή τους με μικρά φορτηγάκια, με βανάκια, κάποιος το διάβασε με εξονυχιστική προσοχή. Διότι ούτε καν στην έκθεση δεν υπάρχει και εδώ πραγματικά έχουμε έλλειψη δεδομένων. Όλοι θέλουμε περισσότερα από αυτά που υπάρχουν. Εάν έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την διόγκωσή του, το νέο σύστημα διοδίων στο Βέλγιο δεν είναι σαφές, δεν είναι μετρήσιμο ακόμα το στοιχείο αυτό. Ακόμα τα στοιχεία πρέπει να τα συγκεντρώσουμε. Οι στατιστικολόγοι των χωρών μας βάλαν πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους αφού συναντηθούν για να ορίσουν τι είναι το minivan, πώς θα μετρώνται αυτές οι μεταφορές και ούτε καθεξής. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι πρέπει να υπάρξει εξακολούθηση στη μελέτη να δούμε τι γίνεται για την υπόλοιπη Ευρώπη επίσης και ίσως να πρέπει να τεθεί και στη Eurostat. Δεν νομίζω η απάντηση αυτή να σας ενθουσίασε, αλλά έχει μέλλον για να καθορίσουμε τι είναι αυτά τα δανάκια. Μιλήσατε για εναλλακτικά καύσιμα και ρωτήστε τι κάνει η Μπενελούξ ε, προς το σκοπό αυτό. Στη μελέτη. Δεν αναφέρεται άμεσα στη μελέτη αυτό, αλλά ξεκαθαρίζεται ότι ναι, διαφέρει η βιωσιμότητα και η εφορία των ε, στόλων να αυξηθεί για να φτάσουμε στους στόχους για το διοξίδιο του άνθρακα. Βέβαια, από πέρσι υπάρχει σύσταση Μπενελούξ για το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων στα πλαίσια της οδηγίας για το κλίμα και τα όσα ορίζει η Ευρώπη. Τα κράτη θα πρέπει να καταθέσουν επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα δράσης τον Νοέμβριο μάλιστα για το πώς θα είναι η σταθμή εκφόρτωσης, ε, ποιος θα είναι ο στόλος, τα οχήματα, τα φορτηγά και πώς θα, κυκλοφορούν τα επόμενα χρόνια. Ως Benelux εμείς έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία και μια δήλωση ε, εκδώσαμε το 2015 που λέγαμε ότι εάν αυτά τα προγράμματα δράση, όταν έρθουν μάλλον με το καλό, που τα συζητάμε εμείς ε, στα Υπουργεία μας, είναι σε πολύ στενή επαφή και ε, υλοποιηθούν, για μας είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι δεν θα έχουμε ένα σταθμό εκφόρτωση ε, από κάθε πλευρά των συνόρων. Ε, θα δούμε πώς θα γίνει με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Ή σε σταθμούς, ε, μάλλον πρατήρια καυσίμων, όχι μόνο για την εκφόρτωση. Θα πρέπει να δούμε στα νέα καύσιμα τι θα κάνουμε και έχουμε και την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα διάδρομο με ασφάλεια σχεδιασμού και για τους ε, μεταφορείς αλλά και για τους διαχειριστές των δικτύων. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό ε, από την οδηγία του κλίματος για τις μεταφορές. Αλλά βεβαίως εργαζόμαστε σκληρά εκεί. Απλώς να προσθέσω με το μικρόφωνο πρώτα. Ε, ρωτήσατε για τις υποδομές τέθηκε η ερώτηση του κυρίου Ρικέ με την, ε, για την διασύνδεση με το βορρά της Γαλλίας. Νομίζω το πλέον σημαντικό έργο αυτή τη στιγμή είναι το νέο κανάλι στο Τένουιζεν για τη διασύνδεση Βελγίου-Γαλλίας τέλο πάντων ίσως κατ' επέκταση και κάτω χωρών, ε, αρκετά εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Όταν ξεκινήσουν, μάλλον τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν και με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση πόσο σημαντικό είναι. Πρώτο βήμα για να ενώσουμε το Ρότερνταμ και το βορρά τη Γαλλία. Έχει ακόμα μέλλον. Αλλά οι αρχίζουν να φτιάχνονται. Και αυτό που βλέπουμε, και το βλέπω και σε σχέση με το δικό σα ερώτημα, είναι ότι για να λύσουμε τοπικά προβλήματα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο σφαιρικά. Όπω αυτό που είπατε για τη διασύνδεση με το Στρασβούργο. Για μα, εντάξει, εγώ Βέλγο είμαι, αλλά μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου δεν είναι καλή η συνδεδομική σύνδεση. Και, έχει κοστίσει και θα κοστίσει και πολλά. Πρέπει λοιπόν να το λύσει κανεί αυτό. Ε, να το λύσει μεταξύ γειτόνων. Μα είναι σοβαρό πρόβλημα. Ναι, αλλά θα κοστίσει πολλά. Και υπάρχει και το θέμα τη πολιτική βούληση. Αλλά είναι και θέμα γεωγραφική ε, προτεραιότητα και θέση. Δεν θέλω εδώ να προσπιστώ του πολιτικού συνέδρου του Βελγίου. Αλλά για τα διεθνή προγράμματα υπάρχουν επενδύσει. Εντάξει. Πρέπει όμω κανεί να ασχοληθεί και με τη συντήρηση του εθνικού του δικτύου. Είναι κάτι που είναι πολιτική επιλογή. Και αυτό τίθεται κάθε φορά. Όπως το είπατε. Όμως χάρη σε αυτή την σε τη συνεργασία να τον κανάλι το Τερνέζεν Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ γειτόνων. Και μετά για τα βανάκια, για τα ελαφρά οχήματα. Πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί υπάρχει πραγματικά μια τάση να αλλάξει ο τύπος φορτηγών που χρησιμοποιούνται από τα βαρέα στα μικρά ε, φορτηγά και αυτά τα βανάκια, γιατί δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τι ίδιε απαιτήσει, δεν έχει απαιτήσει νομοθεσία ούτε τα ίδια για τα έργα κυκλοφορία. Υπάρχει λοιπόν μετατόπιση τρόπου, τροπική στις μεταφορές. Και επίσης, για να το μελετήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να στραφεί και η προσοχή μας. Τώρα ο που ζήτησε πρώτος το λόγο και μετά εσύ. Κανονικά έχουμε τελειώσει, αλλά είμαι και νεόδωρο και μετά θα πάρω και εγώ το λόγο και οι τρει μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μεγάλη ψυχία σας. Ε, εγώ ρώτησα για τις δεξιότητες και τα προσόντα ε, των εργαζομένων. Στην έκθεσή σα επίσης είδα ότι ε, μιλάτε για ψηφιακές φορτωτικές, για πλούσευση των εγγράφων δηλαδή που πρέπει να έχουν μαζί τους ε, η οδηγία των φορτηγών. Ο κύριος Βαντεκρά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για αυτά τα μεγαθύρια, τα φορτηγά. Στο Λουξεμβούργο επιτρέπονται τέτοια. Και στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία επιτρέπονται γιατί τη ότι πάνω από 60% των ε, ομόσπονδων κρατηδίων ε, κυκλοφορούν ήδη. Επιτρέπεται. Δύο σκέλη έχει ερώτηση. Τι γίνεται με το Λουξεμβούργο και τι γίνεται με τη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Ευχαριστώ. Και ο πρόεδρος, μπορώ να σου πω, στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία απαγορεύονται. Στην Πενελούξ και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το είχαμε πει, προσέκρουσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι διασυνοριακό. Ε, ε, ε, ο Κάλλας προσπάθησε να το περάσει, εμείς αντιταχθήκαμε και υπήρξε πλειοψηφία και το σταματήσαμε. Αλλά οι χώρες γιατί είναι τόσο μάγκες και τόσο πονηροί και βλέπω μπροστά μου δύο τέτοιους τύπους, ε, ε, συμφώνησαν σε μια συμφωνία Benelux ε, που υπήρχε η συνθήκη πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα και το επέτρεψαν για αυτά τα τρία κράτη τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία δεν μπαίνουν. Υπάρχουν άλλα κρατήδια που τα επιτρέπουν. Πάντως στο δικό μας κρατήδιο όχι. Δεν, δεν θα πέρασουν. έχω άλλη ερώτηση τώρα εγώ για το ε, σύστημα των διοδίων. Εγώ πάντα φέρνω ως παράδειγμα στην Ελβετία. Αυτό μπορούν να το κάνουν γιατί δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς βάλαμε για τα φορτηγά διόδιο, τέλη δηλαδή, ε, σε όλα ε, τα φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους. Για να μην φεύγουν από τους αυτοκινητοδρόμους να πηγαίνουν σε εθνικές οδούς κτλ. Στην Ισπανία είδαμε ότι έχουμε ένα νέο ε, αυτοκινητόδρομο με κοινοτική συγχρηματοδότηση κτλ. Και, και περνούσε ένα φορτηγό κάθε μισή ώρα. Και πάμε και στην παλιά εθνική οδό και γίνεται χαμό από φορτηγά εκεί πέρα γιατί δεν πληρώνουν, είναι πιο φθηνά. Ε, άμα το κάνεις για όλους τους δρόμους όμως δεν θα πάνε από τον ένα δρόμο στον άλλο. Καταλαβαίνω με τη, σχέση, με τη διασύνδεση Βρυξέλλες-Στρασβούργο ε, ότι είναι ακριβή, αλλά και 900 εκατομμύρια, εντάξει, αλλά τα 800 μέτρα από τη Βαλανσιέν στη και τα χορτάρια στο, στις ράγες. Τι φταίει και τι φταίει, γιατί δεν γίνεται αυτό. 800 μέτρα και κερδίζεις μία ώρα Αβρυξέλλες Βαλανσιέν ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό συνδέροδρομο. Είναι και προσβολή για τον οργανισμό και για την πόλη της Βαλανσιέν. Δεν ξέρω ποιος ήταν παλιά εκεί δήμαρχος. Ε, αλλά τα 800 μέτρα, ε, δηλαδή έλεος. Δεν θα μπορούσατε να μου απαντήσετε, παρακαλώ. Α, και άλλη ερώτηση του Ρικέ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να προσθέσω κάτι. Είναι η πρώτη διεθνής θηρομική ε, γραμμή του κόσμου. Βρυξέλλες Παρίσι περνούσε από εκεί. Ναι, υπάρχουν 800 μέτρα τα οποία αρκεί να ξαναφτιαχτούν η γαλλική πλευρά χρηματοδότη εν μέρη, αλλά ένα εκατομμύριο ευρώ δεν έχει εξευρεθεί από πλευρά Βελγίου. Λίγο απίστευτο. Πιστεύω ότι αυτά τα 400 μέτρα θα επιτρέψουν αυτή την καοδο απο από βορρά-νότο, δίχως να περάσουν από το Παρίσι, το οποίο έχει τεράστια συμφόρηση. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Να προβοκάρω τώρα εγώ. Ένα εκατομμύριο είναι πολλά λεφτά, αλλά 900 εντάξει, κανένα πρόβλημα. Για τώρα, απαντήστε τώρα εσείς. Αυτό το θέμα δεν έχει συζητηθεί στο πλαίσιο του Μπενελούξ αυτό το. Αλλά είπα ότι σήμερα το πρωί μια συνεδρίαση με τον κύριο Μπέλο, του το Υπουργείο Μεταφορών, τον Διευθυντή και θα μεταφέρουμε τα σχόλιά σας, τις ανησυχίες σας που ακούσαμε στο Κοινοβούλιο και αυτή νομίζω ότι θα είναι μια λύση γρήγορη, όχι, όχι δαπανηρή. Θα μεταφέρω λοιπόν αυτά που είπατε. Να φτάσει ό,τι αφορά. Θα, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σας το διαβεβαιώνω. Ένα άλλο στοιχείο και μετά θα δώσω το λόγο στον ε, Γιάννη Μούλεμαν σε ό,τι αφορά τι ε, επαγγελματικέ ειδικότητε. Ε, εδώ και δύο χρόνια συζητιέται και το οποίο χειριζόμαστε εμείς. Χειριζόμαστε εμείς. Δεν είναι μια απάντηση ουσιαστική, αλλά από πέρυσι έχουμε μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την εμβέα αναγνώριση των πτυχίων μάστερ στις κάτω ε, στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο κλπ. Σήμερα λοιπόν θα το ελέγξουμε και σε επίπεδο ε, των μεταφορών και θα δούμε τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο επίπεδο Benelux στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι η προσθέμενη αξία για μας. υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο περί επαγγελματικών προσόντων αλλά σε θέματα μεταφορών υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Όλα αυτά αφορούν την κινητικότητα της αγορά εργασία. ναι, να προσθέσω σε το θέμα της απασχόλησης του κλάδου, στον κλάδο. Κάθε 10 ε, θέσει εργασία συνδέονται με τα logistics, στην εφοδιαστική. Γι' αυτό λοιπόν ο τομέας θα πρέπει να παραμείνει κατάλληλα οργανωμένος και θεωρώ πως ο εξοικονομισμό είναι απαραίτητος και στον τομέα αυτών. Ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να βοηθήσουν και να καταστήσουν πιο, πιο ρευστές τις ε, μεταφορές είναι η ψηφιοποίηση αυτό το οποίο συμβαίνει για το ε, θέμα της ψηφιοποίησης των εγγράφων ε, τονίστηκε και ακόμα και από κάποιους πρωθυπουργούς αν υπάρχει ένα τομέα όπου η ψηφιοποίηση θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω είναι το τομέα των μεταφορών. Ως εκ τούτου λοιπόν για το επόμενο έτος ε, ξεκινήσαμε κάποιο πιλωτικό, πιλωτικό προγραμματισμό και είτε πρόκειται για φορτηγό, είτε πρόκειται για πλοίο, για όχημα. Ξέρουμε ότι απαιτούνται συχνά πολλά έγγραφα, πολλά χαρτιά και η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει σημαντικά. ειδικά στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών. Θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες συμφωνίες μεταξύ των κρατών προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ψηφιοποίηση. Αυτό θα συμβεί αναφίβολα τα προσοχή έτη. Οι, οι, οι πρωθυπουργοί μας το γνωρίζουν αυτό για τελευταίο σχόλιο για τα μεγάλα αυτά τα φορτηγά μαμούθ. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για τα πιλωτικά προγράμματα. Κατά πόσο δουλεύει καλά, γιατί δεν δουλεύει καλά, για ποιο λόγο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι το παράδειγμα ε, τα λουλούδια τα οποία φορτώνονται στην Λίγη θα πρέπει να μεταφερθούν τάχιστα σε ένα αεροδρόμιο πλησίων μπορεί να επιληθεί από το μεγάλα αυτά φορτηγά, τα τεράστια φορτηγά, τα οποία να κυκλοφορούν βράδυ και να μην δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους. Και υπάρχει πολύ καλή παράδοση στο Μπενελούξ, το οποίο θα φροντίσουμε να μοιραστούμε με τους εταίρους μας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και θα ενημερώσουμε και ο καθένα θα είναι φυσικά ελεύθερο να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν αυτή την ενημέρωση. Έχετε καμία ημερομηνία από θα τελειώσει αυτή η πιλωτική μελέτη. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί δεν ξέρουμε ούτε καν πότε θα αρχίσει. Στη Γερμανία είναι 3, 5, 6, 7 τα πιλωτικά προγράμματα και αν δεν ξέρει πότε τελειώνουν και αυτό είναι άδικο. Είναι και κόλπο και τέχνασμα μαζί. Ελπίζω Μπενελούξ να μην το αντιγράψουνε. Μην αντιγράφετε τέτοια κόλπα. Κύριε Πρόεδρε, προσέξτε. Για οι περιβαλλοντικέ μελέτες πρέπει να διαβάσετε για τα μεγάλα φορτηγά. Βεβαίω θα το κάνω, αλίμονο, αν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Βίλεμς και τον κύριο Μόλεμα για τις παρουσιάσεις σας και για τη συζήτηση. Λίγη και καλή, ε, κουραστική μέρα όμως ήταν σήμερα. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη πρέπει να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο σημείο 21 έχουμε τελειώσει, το 22 έχουμε τώρα διάφορα, δεν έχει κανείς κανένα διάφορο, ούτε βλέπω. Και πάμε στο 23 Εσίους που είναι η ημερομηνία και τόπος επόμενης συνεδρίασης Βρυξέλλες, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 στις 9 ώρα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε και ό,τι επιθυμείτε.